Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι θα καταφτάσουν και άλλοι. Να καλωσορίσω τους δύο συντάχτες της εκθέσεως Global Governance 2025. Λοιπόν, είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση του 2025, ο Ματ Μπάρος από το National Intelligence Council μεγαλύτερη υπηρεσία για συλλογή πληροφοριών τη ΕΠΑ και τον Τζοβάνι Γκρέβι που εργάστηκε για πολλά χρόνια στο European Union Institute for Security Studies στο Παρίσι. Είναι μια ομάδα προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ασχολείται με θέματα ασφαλεία. Κάνει έρευνα για θέματα ασφαλεία και προετοιμάζει αναλύσει και προβλέψει επί του θέματο. Λοιπόν, και συνδράμουν την Βαρόνια Άστον Λοιπόν, η έκθεση σας έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικός. Σας δόθηκε ένα σημείωμα back and note και είναι μια πρωτοβουλία ανευπληγουμένη αυτή που ανελήφθη το 2009 για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ανέλαβαν να εκπονήσουν κοινού προβληματισμούς, θα συμμετείχαν διεθνείς εμπειρογνώμονες ε, που συμμετέχουν και σε τέρους μας σε άλλες χώρες όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης στο μέλλον του Global Governance. Και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ θεωρείται όλο και περισσότερο διεθνείς ε, σχέσει, εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από ότι οι παραδοσιακέ δομέ τη διακυβέρνηση. Και λοιπόν, κατεπηγόντω, χρειάζεται να ξεκινήσει ένα στρατηγικό διάλογο όσον αφορά τι ε, μελλοντικέ αυτέ σχέσει τη διεθνή. Η αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ και των άλλων χωρών, με την Κίνα εν πρώτη στην Ιαπωνία και τις χώρες του κόλπου, Ινδία, Νότια Αφρική, Βραζίλια και Ρωσία είναι κάτι που γίνεται και αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να οδηγήσει σε ακριβέστερη αξιολόγηση ενδεχομένων σεναρίων για την διαμόρφωση της global governance στο μέλλον. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει στο όλο πρόγραμμα από την αρχή μέσω του συναδέλφου του James Ellis ε, που είναι εδώ που είχε την ιδέα να προτείνει αυτή την πρωτοβουλία, την κοινή πρωτοβουλία και που δεσμεύτηκε να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Τον ευχαριστώ προσωπικά, τον ευχαριστώ εν ονόματι όλων. Λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη εγώ θα ακολουθούσα την εξή σειρά. Πρώτα να βάλω στον Ματ Μπάρος και μετά στον Τζοβάνι Γκρέβι και ενδεχομένως μετά στο συνάδελφο Έλλης αν θέλει να πάρει το λόγο. Και μετά βεβαίως θα υπάρξει περιθώριο για υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεων. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Κύριε Μπάρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω και να μιλήσω για αυτή την έκθεση που από κοινού ετοιμάστηκε μεταξύ του Εθνικού Συμβουλίου Συλλογής Πληροφοριών, εκεί που εργάζομαι εγώ, και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να αναφερθώ επολίγων στο ιστορικό της εκθέσεως και μετά να σας δώσω κάποια γενική εικόνα των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε. Μετά ο Τζοβάνι μπορεί να επισέθει σε κάποιες επτομέρειες της έκθεσης πριν διεξαχθεί μια συζήτηση επί του θέματος. Ποιο είναι το ιστορικό λοιπόν. Το National Intelligence Council των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε τέσσερα χρόνια ετοιμάζει μια έκθεση για τις παγκόσμιες τάσεις. Ε, εξετάζει μια περίοδο 15 ετίας, 20 ετίας. Η τελευταία είχε δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2008 και την παρουσιάσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αφού δημοσιεύτηκε γιατί κάναμε τη δημοσίευση. Θέλαμε να βοηθήσουμε την επόμενη Αμερικανική κυβέρνηση να προβλέψει τι θα γίνει στα 15-20 χρόνια. Να βοηθήσουμε λοιπόν την κυβέρνηση με τις προσπάθειές της ε, για την ε, κατάρτιση στρατηγικών, όχι μόνο μακροπροθέσμος, αλλά και μέσω βραχυπρόθεσμα. Ένα από τα πορίσματα της εκθέσεως ήταν ότι αντιμετωπίζαμε ένα έλλειμμα διακυβερνήσεως για τις επόμενες ε, δεκαετίες και υπήρχαν διάφοροι λόγοι ε, γι' αυτό και δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες αλλά διεφαίνεται ότι η διακυβέρνηση ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να εξεταστεί ε, περαιτέρω και έπρεπε να δούμε και ποιες δυνατότητες υπήρχαν για αλλαγές όσον αφορά το έλλειμμα της διακυβέρνησης. Όπως ίσως πει και ο Τζοβάνι, ο φορέας του και αυτός κάνει μακροπρόθεσμες μελέτες και κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Προφανώς είναι λογικότατο κατά την άποψή μου οι Ηνωμένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δοθέντων των ρόλων μας δηλαδή που δημιουργούμε και ασκούμε την παγκόσμια κυβέρνηση μέσω των θεσμών που διαθέτουμε θα πρέπει να συνεργαστούμε, να προβληματιστούμε, να δούμε ποιες αλλαγές απαιτούνται στο μέλλον, ε, τι συνέπειες ε, έχει αυτό το έλλειμμα που προανέφερα. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών, η συνάθρηση των προσπαθειών και των πόρων μας οδήγησε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος. Δηλαδή επισκεφθήκαμε κάθε σημαντικό κέντρο ισχύω στον κόσμο για να καταλάβουμε πώς βλέπουν αυτοί τα θέματα της ε, διακυβέρνησης και να καταλάβουμε πού έβλεπαν, ε, ποιε τάσεις διαπίστωναν ότι υπάρχουν. Όπως αναφέρεται από τον τίτλο, ότι είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμιο η παγκόσμια κυβέρνηση, αυτό αναφέρει ο τίτλος, Ποια ήταν βασική ανησυχία, όπως και σε πρώτερες εκθέσεις, ότι για διάφορους λόγους οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι περιφερειακοί θεσμοί που γνωρίζουμε δεν αρκούν όσον αφορά τις τάσεις που διαμορφώνονται. Και υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι ε, που μας οδήγησε αυτό το συμπέρασμα. Πρώτος λόγος. Είδαμε ποιες προκλήσεις μας περιμένουν. Προφανώς τα συστήματα διακυβερνήσεως, αυτά που, το σύστημα που γνωρίσαμε το 1945 και πέρα, ήταν αρκετά επιτυχές Μπορεί να το πει κανείς αυτό, αλλά οι μελλοντικές προκλήσεις, και αναφέρουμε αρκετές, συγκεκριμένα στην έκθεση, που αφορούν τους πόρους, νερό, τροφή, ενέργεια. Οι προκλήσεις αυτές, λέγω, αφορούν και τις συγκρούσεις, χώρες που έχουν μείνει πίσω, που δεν μπορούν οι χώρες αυτές να αναπτυχθούν με τους ίδιους ρυθμούς όπως ο υπόλοιπος κόσμος και άλλα ζητήματα που είναι στον ορίζοντα. Μετανάστευση, αυξανόμενο πρόβλημα. Επανάσταση στη βιοτεχνολογία διάφοροι θεσμοί διακυβέρνησης προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις τάσεις και τις προκλήσεις, αλλά ανεπιτυχώς. Χρειάστηκε λοιπόν να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή είναι μια ομάδα θεμάτων, δηλαδή αυτές είναι οι προκλήσεις, που οι προκλήσεις είναι προϊόντα της παγκοσμιοποίησεως, της μεγαλύτερης αλληλεξαρτήσεως, που είναι κυρίως κάτι εποφελές, έχει θετικά αποτελέσματα για όλους. Βλέπουμε την αυξανόμενη ευμάρεια στον κόσμο, αλλά υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση και δημιουργούνται τα θέματα που προανέφερα. Και λόγω της αλληλεξάρτησης χρειάζεται μια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή ήταν μια ομάδα ανησυχιών. Μετά έχουμε πολυπολικότητα που αυξάνεται στον κόσμο και τα ταξίδια ήταν άκρως διαφωτιστικά στον αφορά αυτό το θέμα. Ταξιδεύοντας και πηγαίνω σε διάφορες χώρες που ανέφερε ο Πρόεδρος και δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες τώρα. Λοιπόν, πηγαίνω σε αυτές τις χώρες μαζέψαν πληροφορίε όσον αφορά το τι γίνεται για την παγκόσμια διακυβέρνηση και πώς το βλέπουν αυτές οι χώρες το σύστημα διακυβέρνησης είχε σχεδιαστεί για την μεταπολεμική περίοδο, μετά το 1945 και δεν έλαμβανε υπόψη τις νέες χώρες που δημιουργήθηκαν. Τότε δεν υπήρχε άλλη ιδέα για την διοργάνωση της διεθνούς τάξεως. Ε, θεωρήθηκε ότι ο ΙΕ ήταν ένας θεμητός θεσμός που θα τα ρύθμιζε αυτά. Αλλά άνευ μεγάλων μεταρρυθμίσεων με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε το παρόν σύστημα τελικά δεν θα ήταν τόσο αξιόπιστο. Και στις χώρες αυτές έβλεπε κανείς, στις ανατολικές χώρες κυρίως περισσότερο από τις δικές, έβλεπε κανείς ότι τόνιζαν την νομιμότητα πολλές δυτικές χώρες σκεφτόταν περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του συστήματος και ότι είναι πρωταρχικό κριτήριο για τη διακυβέρνηση. Στα ταξίδια μας διαπιστώσαμε ότι εκεί η έμφαση ήταν περισσότερο στην νομιμότητα, στην αξιοπιστία. Λοιπόν, αυτές οι νέες χώρες, οι περισσότερες από αυτές είναι φτωχές χώρες, παρόλο που η Κίνα είναι η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία, έχουν τεράστια επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχουν απόψεις που ανήκουν σε μια χώρα που αναπτύσσεται γρήγορα. Και όταν μάλιστα το μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού είναι σε φοβερή φτώχεια. Είναι πιο ισοστρεφής. Ταυτόχρονα όμως περιμένω αυτές τις μεγάλες ε, αλλαγές στους θεσμούς σε παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία μετά την υποβολή τη εκθέσεω, η πρωτοβουλία για την παγκόσμια διακυβέρνηση θα παραμείνει στα χέρια τη Δύση για την ώρα. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε το θέμα. Το πώ θα αλλάξουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αν θεωρήσουμε όμω ότι το όλο διεθνέ σύστημα θα μπορούσε να υπονομευθεί, έχουμε τέσσερα σενάρια τα οποία περιγράφουμε. Θα τα αναφέρω ακροθυγώς. Πρώτο σενάριο παρούσα τάση την οποία περνάμε κάποια δυσκολία. Θεωρούσαμε ότι είναι πιθανό σενάριο, αλλά δεν θα ήταν βιώσιμο λόγω των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Θεμάτων που αναφέρουμε στην έκθεση. Δεύτερο εξίσου πιθανό σενάριο ήταν ο κατακαιρματισμός, ήδη συνέβη αυτό, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, η ύφεση στην παγκοσμιοποίηση οι ρυθμοί της ανάπτυξης πολύ πιο χαμηλή, περιφερειακή προσέγγιση στην ανάπτυξη, δεν είναι καλό σημάδι μακροπρόθεσμα. Θα σήμαινε υπονόμευση του παγκοσμίου συστήματος. Τρίτο σενάριο, το θετικό. Ε, ένα σχέδιο για παγκόσμια διακυβέρνηση το οποίο θεωρήσαμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκτός αν είναι μια, συμβεί με τεράστια κρίση η οποία να οδηγήσει σε συνεργασία και συνεννόηση και όλοι μαζί να ενωθούν. Δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Και τέλος έχουμε τις συγκρούσεις, τη σύγκρουση. Αυτό δεν μπορούμε να το απορρίψουμε, φέρεται απίθανο σε αυτή τη φάση, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ότι και σε, στο παρελθόν η παγκοσμιοποίηση είχε αποτύχει. Άρα δεν είναι εντελώς απίθανο να έχουμε ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα και για αυτή την προσπάθεια παγκοσμιοποίησης που μέχρι τώρα ήταν θετικότατη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας. Θα σταματήσω εδώ, ούτω ώστε ο Τζοβάνι να επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ε, έκθεση. Έχετε το λόγο, Τζοβάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ για να σας δώσω μερικές πληροφορίες για τα πορίσματα, ορισμένα πορίσματα της έκθεσής, μου, της έκθεσής μας. Θα ήθελα να σας παραπέμψω καταρχήν στο έγγραφο που προηγήθηκε αυτό το εγχείρηματος για το νέο παγκόσμιο παζλ 2025 δημοσιεύθηκε το 2006 μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο και είναι πολύ έγκυρο, εξακολουθεί να είναι έγκυρο αυτό το έγγραφο που έγινε στι ΗΠΑ και το βασικό του συμπέρασμα είναι ότι στα πλαίσια αυτών των ιστορικών τάσεων που αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο σύστημα, το συνολικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση και στον προσδιορισμό της μελλοντική ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σταθερότητα της ευρύτερη περιοχής. Και από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες ε, δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν το διεθνές σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει μια επιλογή για το κατά πώς θα αντέξει σε αυτές τις αλλαγές ε, θα γίνει απαθητικό αντικείμενο των αλλαγών ή αν θα συμμετέχει ενεργά θα είναι υποκείμενο των αλλαγών. Αυτό ήταν το βασικό πόρισμα αυτής της έκθεσης που δημοσιεύθηκε το 2006 και νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί αυτό το συμπέρασμα τα τελευταία χρόνια. Γιατί για να είναι κανεί ε, σημαντικός, ε, σημαντικός φορέας αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να γνωρίζει τα συμφέροντά του και τους στόχους του. Και ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φυσικά η εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού πολυμερού συστήματος και φυσικά θεσμικών οργάνων που θα μπορέσουν να, να αντιμετωπίσουν αυτή την αλληλεξάρτηση. Και ήταν και μια φυσιολογική επιλογή του UISS με τους εταίρους μας στην ε, Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούμε στο θέμα της παγκόσμιας διακυβέρνηση και η έκθεση αυτή «Παγκόσμια διακυβέρνηση 2025» εξετάζει το ζήτημα και μέσο και μακροπρόθεσμα και εξετάζουμε με τους παγκόσμιους εταίρους μας ποιο θα είναι το μελλοντικό πλαίσιο της ε, συνεργασίας εν ώψη των ε, προκλήσεων που ανακύπτουν και στη συνεργασία μας με τις αναδυόμενες οικονομίες και δυνάμεις. Από ό,τι φαίνεται δεν πλησιάζουμε σε μία ρηξικέλευθη αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος. Υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι και προτεραιότητα και η κοινή διάγνωση ισχύει για τις βασικές προκλήσεις τις κλιματικές αλλαγές, για παράδειγμα την ευπάθεια ορισμένων χωρών κτλ. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την ομοιοποίηση κάποιων θεσμικών οργάνων. Οπότε ο πολιτικός χώρος, το πολιτικό κλίμα δεν είναι ακόμη πρόσφορο για μια ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση της προηγούμενης πολυμερούς δομής, αλλά στις συζητήσεις διαβλέπουμε κάποιους ενδιαφέροντες, ε, κάποιους ενδιαφέροντες δείκτες σε ό,τι αφορά την μελλοντική πρόοδο και τις εξελίξεις στα θέματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Θα αναφερθώ εν συντομία σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά τον αναδυόμενο ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση κάποιων άτυπων λεσχών, κάποιων άτυπο, άτυπων ομίλων, αυτά τα G που λέμε, το G20 για παράδειγμα, που είναι την τελευταία διετία το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ομίλου, αλλά δεν είναι το μόνο G ή δεν είναι μόνο η μόνη λέσχη που αρχίζει και φαίνεται. Για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα είχαμε άλλη ομάδα χωρών την Βραζιλία, την Νότια Αφρική και την ε, Κίνα. Είχαμε τους BRICS που έδωσαν έμφαση στα οικονομικά ζητήματα. Είχαμε την ομάδα Ήψα από τις νότιες χώρες Βραζιλία, Νότια Αφρική και ούτω καθεξής. Και ενώ οι αναδυόμενες οικονομίες ε, προσπαθούν να κρατήσουν ζηλότυπα την κυριαρχία τους στα πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ανακοινούνται και οι ανάγκες για περισσότερες δεσμεύσεις. Και αυτές οι ανεπίσημες λέσεις ε, οι όμιλοι επιτρέπουν κάποια, κάποιο συντονισμό των πολιτικών στα πλαίσια παγκόσμιων κρίσεων, όπως ήταν η χρηματοπιστωτική του 2008, αφήνοντας όμως ένα περιθώριο λιγμών σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου πρόκειται για ένα σύστημα, μια μορφή διακυβέρνησης που ταιριάζει σε αυτή τη συγκυρία. Εκκληματίζεται στις σημερινές συνθήκες και την αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασία. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αμφισημείς μεταξύ των εταίρων σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα κάποιων δομών, όπως είναι το G20 για παράδειγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις σε ό,τι αφορά το μέλλον του G20. Και μάλιστα λένε θα πρέπει να διαβηρηθεί το πρόγραμμά του, γιατί πριν από δύο χρόνια στόχος ήταν η καταπολέμηση, ο περιορισμός της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Τώρα αρχίζει και διαφυσβητείται η εντολή του και οι αρμοδιότητες του G20, αλλά και οι προτεραιότητες του προγράμματος του G20 γιατί θεωρείται ως ε, προσανατολισμένο προς τη Δύση. Γιατί βέβαια πολλοί τη χαρακτηρίζουν την κρίση ως βορειοατλαντική οικονομική κρίση σε σχέση με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτό είναι άλλο όμως. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά, την ιδιαιτερότητα του G20 σε σχέση με άλλους ομίλους κρατών είναι ότι αυτή η μορφή διακυβέρνησης και ορισμένων ε, χωρών που έχουν κύριο ρόλο και συνέρχονται προκειμένου να συμβάλλουν με τις συνεισφορές τους στη διαχείριση παγκόσμιων προβλημάτων είναι ένα φαινόμενο που θα βλέπουμε όλο και περισσότερο στο μέλλον. Ένα άλλο ε, επίσης ενδιαφέρον σημείο αφορά τις προοπτικές για μια ευρύτερη διαπεριφερειακή συνεργασία σε σημαντικές περιοχές του κόσμου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Νότια Ασία αλλά και η Νότια Αμερική και η Αφρική είναι αντίστοιχες περιοχές. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι ότι θα ε, διευρυνθεί και θα, διευθυ... Ε, θα εμβαθυνθεί η διαπεριφερειακή ολοκλήρωση τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μια δύσκολη και αρκετά αμφιλεγόμενη διαδικασία. Πάντως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που φαίνεται ότι ενισχύουν τον περιφερειακό διάλογο και τον διαπεριφερειακό συντονισμό. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, κατά τη γνώμη των εταίρων μας και των συνομιλητών μας, φαίνεται ότι διεύρυνε την έννοια της, της, της ότι ο καθένας θα πρέπει να στηρίζεται στον εαυτό του. Δηλαδή, ο καθένας θα πρέπει να είναι ικανός να αυτοπροστατευτεί από παρόμοιες ε, οικονομικές κρίσεις. Να μπορεί κανένας να στηρίζεται στα πόδια του αλλά και στις ε, περιφερειακές ε, αγορές. Αυτό για παράδειγμα στην Νότια Ασία και στην Νότια Αμερική. Επίση υπάρχει και μία μετάθεση της εξουσίας σε περιφερειακό επίπεδο. Χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία προσδιορίζουν κατά κάποιο τρόπο το, την κατεύθυνση του περιφερειακού διαλόγου και φαίνεται ότι το κάνουν. Βέβαια, το τοπίο είναι αρκετά πολυσύνθετο και εικόνα περίπλοκη και μερικές φορές και αντιφατική, αλλά το βλέπουμε στις επενδύσεις σε πλατφόρμες ε, διαπεριφερειακού διαλόγου. Αυτές οι πιο ισχυρές χώρες προσπαθούν ε, να, δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και να δρομολογήσουν το διάλογο προς τα θέματα που τους ενδιαφέρει. Βέβαια υπάρχει σύγκληση σε ό,τι αφορά ανάγκη μεγαλύτερου διαπεριφερειακού συντονισμού. Και η Ιαπωνία, για παράδειγμα, αρχίζει και στρέφεται προς τα δυτικά, δηλαδή προς την Ασιατική Ήπειρο και να συνεργαστεί περισσότερο με άλλες ασιατικές χώρες. Αυτός προς το δεύτερο σημείο. Δεν έχω και πολύ χρόνο, γι' αυτό δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Θα περάσω στο τρίτο θέμα. Το, ο τρίτος τομέας καινοτομία και προόδου που υπογραμμίσαμε στην έκθεση είναι ο ρόλος των μη κρατικών φορέων του επιχειρησιακού κύκλου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και επιστημονική κοινότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμβολή και ο ρόλος αυτών των μη κρατικών φορέων θα είναι πολύ πιο σημαντική στην διαχείριση κοινών προκλήσεων από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι μη κρατικοί φορείς συνέβαλαν στη διαμόρφωση του προγράμματος εργασιών και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο χαρακτηριστικό παράδειγμα και βοηθούν και στην εφαρμογή των λύσεων αυτή η μικρατική κρατική Και αν λάβει κανείς υπόψη την περιπλοκότητα, ακόμη και την επιστημονική, την ανάγκη ειδική γνώσης για πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τις κλιματικές αλλαγές για παράδειγμα, το θέμα της παγκόσμιας υγείας, άλλο παράδειγμα, η βιοτεχνολογία, είναι ένα νέο σύνορο της τεχνολογικής πρόοδου, θέλετε, και της των απαιτήσεων για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αν δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, οι κοινότητε τεχνογνωσία, οι επιχειρηματικοί κύκλοι θα πρέπει να συντονιστούν για να καταλήξουν σε προδιαγραφέ και κώδικες συμπεριφορά για τα θέματα αυτά. Soft law, για παράδειγμα, διεθνεί συμφωνίες με τη συμβολή και του ιδιωτικού κλάδου που θα προσφέρει τη γνώση και που θα δώσει θα προσφέρει και ένα βαθμό συμβατότητας των μέτρων ε, και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί τα διεθνή πολυμερή συστήματα μερικές φορές το hard low, δεν είναι δυνατά σε ορισμένες περιπτώσεις, οπότε απαιτείται soft low. Αυτοί είναι οι τρεις τομείς προόδου που φαίνονται να είναι πολλά υποσχόμενοι έτσι, αυτό προέκυψε από τη συζήτηση με του εταίρου μα. Η εκτίμησή μα είναι ότι η πρόοδο σε αυτού του τομεί είναι ευπρόσδεκτη και ενδιαφέρουσα. Δεν υποκαθιστά κατά ανάγκη την ανάγκη πιο ρηξικέλεθης μεταρρύθμιση ε, της παγκόσμια μεταρρύθμιση και των προηγούμενων πολυμερών ε, οργανισμών ή θεσμών, ξεκινώντα από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν όμως ε, όρια για την αναδιαμόρφωση η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πάντως μας έφερε πολύ κοντά στο χείλος του γκρεμού. Το G20 μας βοήθησε να υποχωρήσουμε λίγο από αυτό το χείλος, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά θα έρθουν και άλλες κρίσεις, εξαιτία των κλιματικών αλλαγών για παράδειγμα, και θα χρειαστούμε ισχυρότερους θεσμούς και οργανώσεις, αν μη τι άλλο για την νομιμοποίηση, για το αίσθημα της ιδιοκτησίας και της αντιπροσωπευτικότητας που είναι ένα αίτημα και των ε, αναδυόμενων εταίρων μας. Πάντως, έτσι με αυτήν την πρόοδο μπορούμε να διαβλέψουμε κάποια, κάποιο τρόπο για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Ποιος θέλει να μιλήσει. Ίσως ο συνάδελφος James Ellis θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Να εκφράσω καταρχάς την ευγνωμοσύνη μου στους ε, συγγραφείς ε, της έκθεσης αυτής που κατάφεραν με ευανάγνωστο τρόπο να παρουσιάσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να εξαγάγουν κάποια συμπεράσματα, το οποίο συχνά δεν το βλέπουμε σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να πραγματικά να πληροφορηθούμε μέσω του εγγράφου αυτού. Είναι η πρώτη φορά που το Εθνικό Γραφείο κατήρτισε μια έρευνα με μια υπηρεσία εκτός είπα. Γι' αυτό θεωρώ την ιστορική στιγμή αυτή. Κατά δεύτερον, ήταν ενδιαφέρον το ότι είδαμε ότι στην Κίνα, την Ιαπωνία, στην Ινδία κανείς δεν ρώτησε τι έκαναν από κοινού η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουν τις χώρες αυτές. Η πιο συχνή ερώτηση ήταν γιατί αργήσατε τόσο. Και στην τελευταία μου παρατηρήση είπα ότι το θέμα δεν είναι τόσο να προβλέψουμε το μέλλον. Είναι να παρατηρήσουμε κάποιες τάσεις, να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση προκειμένου να προσαρμόσουμε και την πολιτική μας βάσει των προβλέψιμων συμπερασμάτων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Εξετάζοντας λοιπόν τα θέματα οικονομικής ε, αλληλεξάρτησης ή αν θέλετε του χαρακτήρα αλληλοσύνδεσης των προκλήσεων και το πώς ε, η επιθυμία συνεργασίας αντίκειται πολλές φορές με τις ε, ενστάσεις των εθνικών αρχών Νομίζω ότι καταλήγουμε σε τρία συμπεράσματα. Ότι μιλάμε για έναν πολικό κόσμο, ότι θα υπάρξει ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, ε, μη κρατικών φορέων. Πρώτο συμπέρασμα, όπως ε, καθότι δημιουργήθηκε η Υπηρεσία εξωτερική δράση θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αντιστοιχία με την Εθνική Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών για να υπάρχει αντίστοιχο σώμα και από τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες ε, έκτακτες ε, αποφάσεις που ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε κατά δεύτερον, δεύτερο συμπέρασμα. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια ε, υπενθύμηση της ανάγκης πιο έντονη συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ. ΕΕ. Θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία. Υπάρχει μια στρατηγική αντίληψη για τον ΝΑΤΟ. Υπάρχει και μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Δεν υπάρχει όμως στρατηγική προσέγγιση για τον διάλογο και την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ. Αλλιώς η ατζέντα θα διευρύνεται, ενώ δεν θα ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες. Και τέλος... ότι πιστεύω ότι κύριε Πρόεδρε πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας, γιατί άπτεται διαφόρων πτυχών που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ενημερώσουμε και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους αλλά και τους νομοθέτες σχετικά με τη σημασία του εγγράφου αυτού. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό το στάδιο δίνω το λόγο στο συνάδελφο κύριο Άτκινς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κατά κάποιο τρόπο είμαι απογοητευμένος γιατί δεν είναι πολύ αριθμοί συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα για να εκτιμήσουν το περιεχόμενο του εγγράφου. Δεν το διάβασα ακόμη, αλλά ξέρω φυσικά αρκετά τον συνάδελφο James Ellis για να ξέρω ότι είναι πραγματικά πολύ δεσμευμένος και τα συμπεράσματά του είναι σωστά. Αυτό που έκανα είναι να διαβάσω την ε, σύνοψη και φυσικά άκουσα και αυτά που είπαν οι προσκεκλημένοι μας. Ένα-δύο σύντομα συμπεράσματα. Και μία απλή ερώτηση, η οποία προκύπτει από αυτά. Η εξή. Αν αποδεχτούμε, έστω ότι είμαστε απεσιόδοξοι και όχι αισιόδοξοι, αν αποδεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει στον κόσμο όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε, είτε μιλάμε για τη ΣΥΠΑ, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε για την Άπο Ανατολή. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή δεν συμφωνούμε και εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας, κατά το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική ταυτότητα ή να υπάρχουν πολλοί στόχοι από τα κράτη-μέλη. Αν συμφωνήσουμε ότι ο ΙΕ δεν έχει ουσιαστικά ε, δύναμη ή ότι οργανώσεις όπως η Παγκόσμια Οργανώση παγκοσμια οργανωσια ε, ουσιαστικά ε, δεν έχουν δύναμη δράσης Όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι αρκετά δύσκολα και περίπλοκα και επί του παρόντος δεν φαίνεται να προσεγγίζονται. Άρα η έκθεση αυτή καταλήγει στα εξή, στα, παρόμοια συμπεράσματα. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να θέσω είναι αρκετά απλό. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Il collega Dziękuję bardzo. Ευχαριστώ. Παραπονιέστε ότι είναι λίγοι βουλευτές παρόντες. Εγώ προτιμώ λίγοι αλλά εκλεκτοί, λίγοι αλλά που ενδιαφέρονται πραγματικά. Ούκαν το πολλό το έφα όπως ξέρουμε. Δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε αμήχανα ή δυσάρεστα επειδή είναι λίγοι βουλευτές. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο θέμα σε νέο το πρωί προγραμματισμένο, ε, είναι αναμενόμενο να έχουμε τέτοια προσέλευση. Γιατί σε 9 το πρωί δεν έχουμε ακόμη συγκεντρώσει όλες μας τις πνευματικές δυνάμεις για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τέτοια θέματα. Φυσικά πρέπει να διαβάσουμε το κείμενο και θα πρέπει κανείς να έχει άψογη γνώση των Αγγλικών για να κατανοήσει ένα τόσο δύσκολο κείμενο. Γι' αυτό τις παρατηρήσεις μου θα ήθελα να τις εξετάσετε κάπως πιο γενικά, γιατί ελάχιστο χρόνο είχα για να ρίξω μια ματιά. Πάντως, αυτό το εγχείρημα είναι χρήσιμο γιατί δημιουργεί πολλές αμφιβολίες και είναι ενδιαφέρον γιατί πολλές εκθέσεις έχουν πολύ αποστομωτικό χαρακτήρα και κατηγορηματικό. Είναι σημαντικό όμως να υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες που δημιουργείται και να αφήνετε αυτές τις ε, λευκές σελίδες. Είναι σημαντικό νομίζω και πολύ υπεύθυνο για κάποιο διανοούμενο να αφήνει αυτή την αμφιβολία και ουσιαστικά αυτό προκύπτει από την ανάγνωση της έκθεσης. Αυτή η αβεβαιότητα και αυτός ο απρόβλεπτος χαρακτήρας πολλών παραγόντων για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση. Επίσης λέτε ότι οι μη κρατικοί φορείς και παράγοντες θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη επιρροή. Και αυτοί οι μη κρατικοί παράγοντες είναι η επιχειρηματική κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών και αυτό δείχνει πώς ε, προσδιορίζουμε ένα νέο φαινόμενο που δεν ξέρουμε όμως προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά εγώ πιστεύω ότι χωρίς συνέχιση, κάποιο είδους ε, συνέχεια τέτοιου είδους ε, ε, εγχειρήματος θα έχουμε την αίσθηση του κορεσμού. Θα πρέπει λοιπόν να επιχειρήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το κόπο, να κάνουμε την προσπάθεια να εξηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχω τρεις ερωτήσεις και ξέρω ότι δεν το γράψετε αυτό στην έκθεση, αλλά Μπορείτε να μου δώσετε μία πιο ε, κατηγορηματική απάντηση. Γιατί, για παράδειγμα, για το σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν το θεωρείτε ένα αποτελεσματικό, θα πρέπει να το πούμε ρητά και κατηγορηματικά. Βλέπουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ και δεκαετίες το προσπαθούμε και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεταρρυθμισής της μας απασχολεί. Δεύτερον, ελάχιστη ε, έμφαση δώσατε στην τεχνολογία. Μιλήστε για τη βιοτεχνολογία και τις πρόοδο της βιοτεχνολογίας, αλλά δείτε τίποτα για το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο έχουμε τεράστια πρόοδο και η επιρροή του διαδικτύου επηρεάζει πολύ σοβαρά και όλα τα άλλα φαινόμενα που αναφέρεται στην έκθεσή της στην έκθεσή σας. Επίσης, ε, λέτε πολύ διακριτικά ότι είναι πιθανές και κάποιες ένοπλες ε, σειράξεις. Αλλά φυσικά και το θέμα των τρομοκρατικών απειλών έχει τεράστια σημασία. Βλέπετε τι συμβαίνει με την, με την κινητικότητα των, ε, ανθρώπων. Υπάρχει μεγάλο θέμα και υπάρχει πιθανότητα ένοπλων σειράξεων όπως το επισημαίνετε, τι είδους πιθανότητα και τι ένοπλε σειράξει έχετε υπόψη. Ευχαριστώ. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να υπογραμμίσουμε ότι η πρωινή συνεδρίαση που καθορίστηκε έτσι 9 σχετίζεται με το γεγονό ότι ο κύριο Μπάρος θα πρέπει να επιστρέψει στη ΣΥΠΑ με το αεροπλάνο το μεσημέρι. Γι' αυτό έγινε το προεύθυνο συνεδρίαση. Η ποιότητα είναι εγγυημένη από τι παρεμβάσει σα. Ακόμα μια φορά ο συνάδελφο Σεβερίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα λιγάκι. Άρα μιλώ με πάσα ταπεινότητα, γιατί δεν έχω ακούσει τις εισαγωγικέ ε, παρουσιάσεις. Αισθάνθηκα υποχρεωμένο ωστόσο να ζητήσω το λόγο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Πράγματι, θεωρώ ότι θα πρέπει να διοργανώσουμε και άλλες συναντήσεις για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά πιο εις βάθος. Να είμαστε πιο εστιασμένοι σε διάφορα θέματα και να προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα επιτρέψτε μου. Προσπαθώντας να φανταστούμε την παγκόσμια διακυβέρνηση και συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε και μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Γιατί θεωρώ ότι δύο ερωτήματα είναι πολύ επίκαιρα. Μπορούμε να διαμορφώσουμε τον κόσμο όπως είναι ή πρέπει να διαμορφώσουμε τον κόσμο όπως θέλουμε. Γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα και Αυτήν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εκ παραλίλου όμω, ενδεχομένως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να πρέπει να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα προκειμένου να οργανώσουμε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ έχω την αίσθηση και σας ερωτώ αν συμφωνείτε ότι μεταξύ των μεγάλων παράγοντων θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ε, νέο ε, αναδυόμενο παράγοντα αλλά τέλο πάντων, μεταξύ των μεγάλων παραγόντων θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πιο μεγάλο δυναμικό αλλαγή και οι αλλαγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το πιο μεγάλο δυναμικό για να επηρεάσουν την παγκόσμια τάξη, την μελλοντική παγκόσμια διακυβέρνηση. Ίσως και να κάνω λάθος, αλλά δεν θεωρώ ότι η Κίνα θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αλλάξει την παγκόσμια τάξη. Δεν θεωρώ ότι ούτε η ΕΠΑ τελείως διαφορετικό παράδειγμα, έχουν δυνατότητα να αλλάξουν το εσωτερικό τους, αλλά και το, την παγκόσμια τάξη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, αν καταφέρουμε να είμαστε πιο ενωμένοι, αν καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική σημασία, τότε μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά πολλά πράγματα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει σήμερα να ορίσουμε κάποια κέντρα, γιατί μιλάτε για μια πολυπολικότητα Ποιοι είναι αυτοί οι πόλοι, πώς μπορούμε να τους ορίσουμε. Μιλάμε για τις κορυφές ε, πυραμίδων, μιλάμε για το ε, ε, κέντρο, το επίκεντρο κάποιων κύκλων, κάποιων δικτύων. Μία άλλη παρατήρηση. Μία πολύ δύσκολη έννοια σήμερα είναι η έννοια της γειτονίας, γιατί από τη στιγμή που θα ξέρουμε ποια θα είναι τα κέντρα θα πρέπει να ορίσουμε και τις περιοχές γειτονίας και κυρίως ε, πρόβλημα που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις ε, κοινής, ε, κοινών περιοχών γειτονίας. Για παράδειγμα, όπως είναι η Ρωσία σήμερα. Έχουμε και κάποιες πιο ακραίες περιοχές γειτονίας, όπως για παράδειγμα η Αφρική, που είναι κοινή περιοχή μεταξύ Ασία και Ευρώπης, ή για παράδειγμα η Λατινική Αμερική, που αποτελεί κοινή περιοχή γειτονίας μεταξύ Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται λοιπόν με τις κοινέ αυτές περιοχές γειτονίας και πώς επηρεάζει αυτό το όραμα της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Για να κλείσω, να αναφέρω ότι θεωρώ ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο μηχανισμό επικουρικότητας. Γιατί, γιατί μιλάμε για την ε, διανομή, την κατανομή ευθυνών. Δεν μιλάμε για ένα μηχανισμό με αντίβαρα αυτόματης ε, ισοστάθμισης. Πώς μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν την επικουρικότητα αυτή και πώς μπορούμε σε έναν πολικό κόσμο να αναζητήσουμε την ισορροπία και όχι την ασυμμετρία. Ίσως να σας βομβάρδισα με ερωτήσεις, αλλά ήθελα απλά να γραφτούν και στα πρακτικά κάποιες τέτοιες παρατηρήσεις, κάποιες τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ο συνάδελφος Κάτσιν. Αν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ και να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους για το υλικό που μας έδωσαν. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ καλής ποιότητας. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι παρουσιάζονται τα εξής διλήμματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβανόμαστε την ε, ανάγκη αλληλεγγύης, στην αλληλεξάρτηση και την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Επίρου και του κόσμου. Και επίσης ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα, μοντέλο για άλλους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η αντίληψη στην Αμερική για τις προκλήσεις αυτές. Οι ΗΠΑ μπορούν να αποτελέσουν λοιπόν υπόδειγμα, μοντέλο για τον κόσμο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προκλήσεων αυτών. Και να σας επιστήσω την προσοχή στην τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση. Η κρίση αυτή με τρόπο πρωτόγνωρο έπληξε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν φοβούμαστε την τρομοκρατία, φοβόμαστε να χάσουμε τη δουλειά μας. Ο ενεργός ε, πληθυσμός, αλλά και οι συνταξιούχοι φοβούνται. Φοβούνται γιατί τις συντάξεις του μέλλοντος. Διαμαρτύρονται στην Ευρώπη ο κόσμος και αυτό καταδεικνύει με τρόπο σαφή τον φόβο που επικρατεί στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας. Δεδομένου λοιπόν ότι γνωρίζουμε τις αιτίε της κρίσης αυτής, ήταν ε, πραγματικά ελλείμματα ολόκληρων δεκαετιών, ελλείμματα τα οποία καλύπτονταν αγοράζοντας ε, ασιατικές ε, αξίες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι οι ΙΠΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για μας ε, στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να μάθουμε από τις ΙΠΑ και πώς μπορούμε από κοινού να ζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Να προσθέσω μία ερώτηση, αν επιτρέπετε. Η global governance, αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε διεθνές επίπεδο και συνεπάγεται τη συνεργασία πολλών φορέων. Χρειάζεται διαχείριση περιπλόκων προβλημάτων. Το νερό, ενέργεια, φερρυπίν, μετανάστευση, συγκρούσεις. Αυτό από τη μια, από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν στατικικά συμφέροντα εθνικά κάποιων μεγάλων χωρών όπως είναι η Κίνα που λειτουργεί εντατικά σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως στην Αφρική για να αποκτήσει φυσικούς πόρους που είναι στρατηγική σημασία για την ανάπτυξή της και όχι μόνο. Το ερώτημά μου λοιπόν το εξή. Ποιο είναι το επίπεδο δυσκολίας που έχετε μπροστά σα όταν προσπαθείτε να συγκεράσετε την απέτηση που υπάρχει για μια παγκόσμια δικυβέρνηση από τη μία και εθνικού εγωισμού από την άλλη, στρατηγική φύσεω. Κυρίω επισηματικότητα των θεμάτων όπω είναι η ενέργεια, και το επαναλαμβάνω αυτό. Απ' την άλλη, δεύτερη ερώτηση. Θέλουμε να εφαρμόσουμε αναπτυξιακά μοντέλα, κυρίως για τις χώρες τις πιο φτωχές. Διαπιστώσατε αν υπάρχει κάποια δυσκολία στο να βρεθεί μια governance σε τοπικό επίπεδο που επιτρέπει αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Γιατί ξέρουμε ότι συχνά τα προγράμματα συνεργασίας δεν καταλήγουν σε αποτελέσματα τόπου για τον τόπιο πληθυσμό, διότι υπάρχουν διάφορες υποδομές, σειρά υποδομών ή μάλλον έλλειψη υποδομών, κάτι που καθιστά αναποτελεσματική την ε, παρέμβαση. Αυτό είναι το ερώτημα το δεύτερο που είχα να θέσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη για αυτές τις ε, ερωτήσεις. Είναι παρόμοια ερωτήματα όπως αυτά που είχαμε υπόψη μας όταν συντάσαμε την έκθεση. Κάτι άλλο βασικό που θέλω να τονίσω. Αυτή η έκθεση, όπως και άλλε που ετοιμάσαμε όσον αφορά τι παγκόσμιε τάσει, είναι μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε μια διαδικασία. Δεν είναι κάτι οριστικό. Και όπως είπε και κάποιος βουλευτής, εδώ δεν έχουμε όσες απαντήσεις θα θέλατε ενδεχομένω και προφανώς είναι πολύ αβέβαιο το μέλλον και επανειλημμένα το αναφέρουμε αυτό. Ελπίζουμε όμως ότι η έκθεση οδηγεί σε συζήτηση και δράση επίση. Ένας από τους βασικούς στόχους που βλέπω να απορρέει από αυτό το προκαταρκτικό εγχείρημα είναι ότι η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται και όσον αφορά την ανάλυση και όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών και όσον αφορά τον προβληματισμό για τα επόμενα βήματα. Και ελπίζουμε ότι αυτό το έγγραφο θα προβάλλει διάφορα θέματα και προκλήσεις και θα δίνει αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τις αναμενόμενες προκλήσεις που θα οδηγήσει σε μια κάποια κίνηση όσον αφορά τον προβληματισμό και από τις δύο πλευρές. Να ξεκινήσει δηλαδή μια διαδικασία για την αντιμετώπιση των απαιτουμένων αλλαγών όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στις απόψεις που έχουμε για την τεχνολογία. Και χαίρομαι που ο κύριος βουλευτής αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Σωστά είπε ότι έχουμε ένα κεφάλαιο για τη βιοτεχνολογία, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και το διαδίκτυο. Και το σημαντικό είναι το εξή. Πώς βλέπουμε το, τη λειτουργία του διεθνού συστήματος στο μέλλον. Το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διευκόλυνση της κοινωνίας των πολιτών, των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και όπως είπε και ο Τζοβάνι στην παρουσίασή του, η κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, η κοινωνία των πολιτών δημιουργεί διασυνδέσεις και τις διευκολύνει. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς το διαδίκτυο. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλο και περισσότερο πληθυσμοί διασυνδέονται και η κοινωνία των πολιτών επεκτείνεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου εκεί υπάρχει κάποια έλλειψη και αυτό θα γίνει ουσιαστικά μέσω της επαναστάσεως της πληροφορικής. Πράγματι, όπως λέτε, η τεχνολογία είναι βασικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων. Θέλω να σχολιάσω το πώς βλέπουμε το μέλλον του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης και στο έγγραφο αναφέρουμε ότι οι επίσημοι θεσμοί χρειάζονται μεταρρύθμιση. Όμως και άλλα βασικά στοιχεία που ανέφερε ο Τζοβάνι, περιφερειακοί θεσμοί, κοινωνία των πολιτών, η G, 20 που είναι ε, ανεπίσημοι θεσμοί, θα έχουν ε, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα και δεν μπορεί κανείς να κινηθεί χωρίς ανεπίσημες δομές. Πρέπει και αυτές να συμμετάσχουν. Και αυτή είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον. Πέρα από τα σημαντικά στοιχεία που είναι η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία, σε 15 χρόνια θα έχουμε και δεύτερο επίπεδο διαφόρων σημαντικών χωρών, όπως είναι η Ινδονησία, τύπου Ινδονησίας, Μεξικού, Κολομβία ε, κλπ. Οπότε έτσι το παγκόσμιο σύστημα θα λειτουργεί όλο και πιο δύσκολα. Και για να λειτουργήσει ο, πολυπολικός κόσμος χρειάζονται πολλές άτυπες δομές που υποστηρίζουν επίσημους θεσμούς που έχουν ομιμότητα κυρίως όσον αφορά τις παρεμβάσεις. Χρειάζεσαι ένα υπόστρωμα, χρειάζεται ένα υπόστρωμα ανεπισήμων θεσμών, ομαδοποίησεων, διαφόρων περιφερειακών ε, οργανώσεων, κοινωνιών των πολιτών, ούτως ώστε να λειτουργήσει το σύστημα. Τζοβάνι. Well, thank you very much, in fact, for Σας ευχαριστώ, ήταν πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις. Δυστυχώς ε, δεν προλαβαίνουμε να τις απαντήσουμε όλες διεξοδικά και να επισέλθουμε σε βάθος όπως θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά το τι μέλη γενέστε, γιατί πολύ ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και το να κρίνουμε κατά πόσο η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι αποτελεσματική ή αναποτελεσματική. Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, άρχισε να φθήνει την τελευταία δεκαετία εξαιτία των νέων ε, ειδών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ε, και εξαιτία της ελεξάρτησής τους. Γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων των παγκόσμιων θεσμών και οργανώσεων, αλλά και υπάρχει και μια περιπλοκή του παγκόσμιου προγράμματος εργασιών, γιατί οι διάφορες δυνάμεις, σχηματισμοί δυνάμεων έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Σίγουρα είναι τεράστιες προκλήσεις για τη νέα δομή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι πλησιάζουμε ένα σημείο καμπής, μια ε, ιστορική στιγμή συνταγματικής αναδιάρθρωσης και άρδιν αναμόρφωσης. Σίγουρα θα χρειαστούμε νέα joint ventures, νέους τρόπους ε, διεξαγωγής της παγκόσμιας συνεργασίας και κάποια, κάποιες ανεπίσημες πτυχές, κάποιες άτυπες πτυχές ή πρακτικές ε, καινοτομίες θα χρησιμοποιηθούν πολύ και περισσότερο. Και υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα, στην παγκόσμια υγεία για παράδειγμα ή στην ε, συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων τον κύκλο των ακαδημαϊκών, των μεγάλων φιλοθροπικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών και υπάρχουν καλά παραδείγματα στα, θέματα ασφάλειας, τροφίμων και ύδατος για παράδειγμα. Υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες σε ψηλό πολιτικό επίπεδο, αλλά με άτυπο τρόπο, για παράδειγμα το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας ή του περιορισμού της διάδοσης των όπλων. Αυτές τις καλές πρακτικές θα προσπαθήσουμε να τις αξιοποιήσουμε και να διασυνδέσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες με το επίσημο πλαίσιο. Που με το επίσημο πλαίσιο που αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί, να, θα χρειαστεί μια μεταρρύθμιση για να αυξήσει και την αποτελεσματικότητά του, αλλά και την νομιμοποίησή του και την προβλεψιμότητα αυτής της συνεργασίας. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές άδικα κατηγορείται ως παρακμάζουσα δύναμη, ως φτύνουσα δύναμη. Εγώ πιστεύω ότι είναι τεράστιο το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για να γίνει μια μόνιμη εξουσία, αλλά και μια ανερχόμενη δύναμη. Και το είδος της λύσης που προσφέρει στη Διεθνή Τράπεζα Διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεισφορά της είναι πολύ έγκυρη κατά τη γνώμη μου και το επισήμανα αυτό και πολλοί εταίροι μας. Αλλά δυστυχώς μερικές φορές ε, δεν έχει πολιτική συνοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλοκαίρι ε, εξαιτία της ε, οικονομικής κρίσης και του ευρώ ουσιαστικά ε, λαβώθηκε η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του ίδιου της του μοντέλου. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες συνταγές που υπάρχουν. Η Κοπεχάγη, για παράδειγμα, είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα που θα μπορούσε να εξεταστεί. Και να ολοκληρώσω την ερώτηση του Προέδρου σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά μοντέλα και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί είναι που θα δούμε την προσέγγιση και των Πολιτειών και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν όμως διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει εδώ να βρούμε κάποιους τρόπους σύγκλησης, κάποιους κοινούς παρανομαστές, ώστε να δούμε πού μπορούμε να συναντηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά χρειάζεται πολιτική διακυβέρνηση για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση. Η Κίνα, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για τη μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και την καλύτερη πολιτική διακυβέρνηση. Είναι σημαντική η διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, αλλά εκεί έγκυται και η πρόκληση να βρούμε τη χρυσή τομή, το κοινό έδαφος, το κράτος δικαίου και τη σταθερότητα που είναι ενδιαφέρον και συμφέρον για όλους και πώς θα μπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να συνεργαστούν με διεθνείς φορείς για την ανάπτυξη κάποιων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα από τους Αφρικανούς εταίρους μας. Ε, πολλό δε μάλλον που αυτοί έχουν ένα σημαντικό έλλειμμα γνώσης Και στην Αφρική, εδώ, οι πρωταγωνιστές και οι κρατικοί και οι μη κρατικοί φορείς ε, διαπιστώνουν ένα μεγάλο έλλειμμα γνώσης, ένα μεγάλο έλλειμμα τεχνολογίας για να υποστηρίξουν τις δικές τους επεμβάσεις. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα για το ρόλο των μη κρατικών φορέων στην παγκόσμια διακυβέρνηση είναι το επιχείρημα της ε, ανισότητας ό,τι αφορά το ρόλο της ε, συμβολής και της παρουσίας μη κρατικών φορέων και του επιχειρηματικού κύκλου και της κοινωνίας των πολιτών. Ένα τμήμα της συζήτησης στο δυτικό κόσμο είναι ότι ε, ακριβώς υπερισχύουν ε, επιχειρήματα του δυτικού κόσμου, αλλά τίθεται να αμφιβόλη δυνατότητα και άλλων μη δυτικών φορέων ε, να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις και να διεκδικήσουν κάποιο είδους ιδιοκτησία Ιδιαίτερα στις, στους αναπτυσσόμενους, στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι πολύ σημαντικό το αίτημα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους σχηματισμούς. Για να απαντήσω στον συνάδελφο Ρόμπερτ Άτκινς για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί η βάση του εγγράφου είναι, αν θέλετε, το ενδιαφέρον που έχουμε προς την Ινδία, προς τη Μόσχα, προς ε, άλλες χώρες. Κάποια στιγμή στο επόμενο έτος, στην Ουάσιγκτον, θα γίνει μια συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, τάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί θα πρέπει να παρίσταται σε τέτοιες συναντήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμορφώνεται ένα, ένα, ένα παγκόσμιο δίκτυο και δεν μπορούμε πλέον να μην συμμετέχουμε σε αυτόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ τους κυρίους συζητητές, τον κύριο Μπάρους και Γκρέβη. Σημαντικό το θέμα και κάποιος έκανε μια, απέθυνη μια πρόσκληση να προτείνουμε στη γραμματεία άλλη μια συνάντηση. Το δέχομαι αυτό. Να έχουμε με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ήσασταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Εξετάζουμε τις τροπολογίες που κατατέθησαν σε αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Πελιού ε, για τη χωρίς εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως για τα δάνεια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύησης. 61-61 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Και το θέμα που κάλυψε ο κύριος Πεγιών είναι σίγουρα σημαντικό και το Κοινοβούλιο σε, στα πίσω συναπόφαση θα τοποθετηθεί. Και μετά τη δημοσίευση της Επιτροπής των Σοφών για την χρηματοδότηση, εξωτερική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, ξεκίνησε η σύνταξη της εκθέσεως. Λοιπόν, πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πεγιόν και μετά θα ακολουθήσουν οι διάφοροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Ήδη έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής μας για την προσπάθεια που έκαναν ε, και τη σοφία που έδειξαν κατά... με την κατάθεση των 60 περίπου τροπολογιών που αναφέρατε και μάλιστα στο στενό χρονικό περιθώριο που είχαμε στη διάθεση μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους βοηθούς που μέχρι αργά το βράδυ χθε ε, με βοήθησαν στην ε, σύνοψη αυτών των ε, τροπολογιών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου, ιδιαίτερα τον κύριο Λάμστορφ και την κυρία Χάουτάλα, γιατί καταφέραμε αυτούς τους συναδέλφους και να εμπλουτίσουμε το κείμενο, αλλά και να καταλήξουμε σε περίπλοκα ζητήματα, σε σημαντικές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ και τη γραμματεία τους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή τους γιατί ήταν πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα. Έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι πριν και η ΕΤΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευτυχώς όταν του ζητούσαμε ε, αντίδραση και σχολιασμό των προτάσεων ε, έσπευσαν αμέσω ε, να μας ικανοποιήσουν. Ελπίζω το σημερινό κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές. Δεν θα επανέλθω στα θέματα που μας απασχόλησαν στις προηγούμενες συζητήσεις. Θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς μερικές τροπολογίες δεν μπορέσαμε να τις ε, συμπεριλάβουμε συμβεστικές τροπολογίες γιατί βρίσκονταν εκτός θέματος ουσιαστικά, εκτός του θέματος της ε, εντολής ή της ανανέωσης εντολής. Γιατί μερικοί ήταν και κατά της ε, ιδέας ε, της εντολής αυτής και του ποσού που αντιπροσωπεύει, που είναι περίπου 2 δις ευρώ. Η άλλη ήταν, κατά της, ήταν υπέρ της κατάργησης των περιφερειακών ανώτατων ορίων εγγύησεων. Επίσης, απορρίψαμε μία τροπολογία για, τα, για για τη μη χρηματοδότηση προγραμμάτων από την ΕΤΕ, σχεδίων που θα οδηγούσαν σε αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2016. Σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες της κυρίας Κοπά, η Επιτροπή μας, όπως και οι υπόλοιπες, ε, ζητήσαμε τακτική ενημέρωση, περιλήφθηκε ε, αυτή η τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία της κυρίας Χαουτάλα για τις εγγύησει που δεν θα έπρεπε να εξάπτουν το κλίμα σε ορισμένες ε, περιοχές. Αυτό το είχαμε πει και στην πρώτη συνεδρίαση και ε, η τροπολογία του κυρίου Χοντή σε ό,τι αφορά τη σημασία των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου κλάδου. Φυσικά δεν μπόρεσα να δεχτώ αυτούσες όλες τις τροπολογίες. Γι' αυτό και προσπάθησα, και ίσως θα είναι λίγο δύσκολο για την αυριανή ψηφοφορία, να συντάξω συμβαστικές τροπολογίες. Πέντε από αυτές δεν δημιουργούν και πρόβλημα και έχουμε και έξι προφορικές τροπολογίες που συντάχθηκαν ως προ... επίσης συμβαστικές. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας δώσω τους αδρούς άξονες αυτών των ε, τροπολογιών. Πολλές τροπολογίες προσπαθούσαν να βελτιώσουν το θέμα της διαφάνειας και της ε, δημοσιότητας ε, των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε αρκετέ τροπολογίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερος άξονας που δεν έγινε αντιληπτό στην αρχή, αλλά τελικά καταφέραμε να τον συμπεριλάβουμε, μία σύγκληση των προσεγγίσεων της BERT, ε, της Τράπεζας Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης και της ΕΤΕ. Ιδιαίτερα για την εξωτερική δράση, αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Και τρίτος άξονας ήταν η εξασφάλιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πέραν της φάσης της ε, έγκρισης ή της επικύρωσης του σχεδίου του προγράμματος, που πολλές φορές γίνεται με πολύ γενικά έγγραφα. Εμείς ε, διεκδικήσαμε το δικαίωμα αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να επεμβαίνει και στην εκτελεστική φάση του προγράμματος, φυσικά όταν υπάρχουν προβλήματα. Και τέταρτος άξονας είναι η στήριξη της, του ανεξάρτητου Συμβουλευτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ΕΤΕ. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως αυτό με αυτή την πρόταση. Έχουν μείνει κάποιες εκκρεμότητες ε, με κάποιο, ορισμένα ζητήματα που είναι τα πιο ακαθόδη. Κάποιοι βουλευτές, όχι ομάδες πολιτικές, αλλά βουλευτές. Και είχαμε αντιληφθεί από την αρχή αυτή τη δυσκολία. Κάποιοι βουλευτές λοιπόν έχουν επιφυλάξει ό,τι αφορά την διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων χωρών, προκειμένου να προσταθούν ακόμη τέσσερις που δεν πρόκειται να κατονομάσω εδώ. Θα ήθελα παρόλα αυτά να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Πρόκειται για ένα σημαντικό ε, θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει, ε, παρά τις αγαθές προθέσεις, να, να στερήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να βοηθήσει και από τους δικαιούχους τη δυνατότητα να λάβουν τη βοήθεια. Άλλωστε νομίζω ότι έχουμε ενισχύσει την ε, πλαίσιο και την οριοθέτηση των επενδύσεων. Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα, ακόμη πιο ισχυρό. Αντιλαμβάνομαι για ποιου λόγου είστε κατά της ε, διεύρυνση, για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Αλλά είναι σημαντικό ο άξονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι η αντίστοιχη ε, διεύρυνση της δυνατότητας επέμβασης της ΕΤΕ, ανάλογα με την παράταση της εντολής, οπότε να διεκδικεί περισσότερα κονδύλια. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε από τη μια να ζητούμε περισσότερα κονδύλια και από την άλλη να καταρρύπτουμε τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της αύξησης. Ελπίζω πάντως να καταλήξουμε τελικά σε μια ικανοποιητική για όλους λύση, που δεν θα διακυβεύει την ε, συνοχή της έκθεσης. Επίσης, ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι μείζονες προσανατολισμοί της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έγιναν δεκτοί σε μεγάλο βαθμό και από τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμού, τον κύριο Κάλφιν βρίσκουμε στην έκθεσή του τους βασικούς προσανατολισμούς και της δικής μας Επιτροπής. Θα πρέπει να μείνουμε συσπηρωμένοι, να στηρίξουμε τις θέσεις μας, να μείνουμε ενωμένοι, φυσικά να κρατήσουμε τη συνεργασία και με τους συναδέλφους των άλλων επιτροπών και φυσικά πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και που προβλέπει διαβουλεύσεις και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Μια χρονοβόρα διαδικασία έχουμε μπροστά μας, Αύριο θα εξετάσουμε και έξι προφορικές τροπολογίες, κάτι που δεν απλουστεύει φυσικά τη διαδικασία της ψηφοφορία, αλλά ελπίζω ότι θα ικανοποιηθούμε όλοι. Ευχαριστώ για το συνεργάσιμο πνεύμα που δείξατε. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή για αυτή την άψογη παρουσίαση και για την εργασία που τον περιμένει. Σκιώδης εισηγητής, ο συνάδελφος ο κ. Λάμστορφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Λειτουργήσαν όλα άψογα και φυσικά, όπως είπαμε, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Οι συνάδελφοι θα λάβουν, θα δουν ότι κάποιες ε, τροπολογίες τις έχω αποσύρει. Ήταν τεχνικό το ζήτημα, αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής. Και θα ήθελα να το ξανασκεφτεί ο εισηγητής σε ό,τι αφορά το παράρτημα 2 σημείο β, παράγραφος 1 και υποπαράγραφος 1. Ακούγεται πάρα πολύ τεχνικό αυτό το θέμα και πάρα πολύ σύνθετο. Να σας εξηγήσω περί τίνες πρόκειται. Στον κατάλογο των χωρών στις οποίες ε, δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Μπορεί να γίνεται αυτό ε, και με την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από μόνη της η τράπεζα, χωρίς να χρειαστεί να διαβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αναφέρονται κάποιες χώρες εδώ, για τις οποίες προβλέπεται μία εξαίρεση. Χώρες για τις οποίες υπάρχει συναπόφαση κατά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι χώρες αυτές οι οποίες ως τώρα συμπεριλαμβάνονταν σε εξαίρεσης Αφγανιστάν, Μπουτάν και Ταϊβάν. Εγώ θα πρότεινα το εξή. Και νομίζω ότι από πλευρά Κοινοβουλίου πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους. Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ε, πολιτικώς ευαίσθητων χωρών και να συμπεριλαμβθεί αυτός ο κατάλογος των χωρών στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες ε, προβλέπεται στην απόφαση, εξαίρεση. Προτείνω λοιπόν τις τροπολογίες 98, 99 και 100 τη Λιβύη, τη Λευκορωσία, την Καμπότζη και την Ιεμένη. Οποιοςδήποτε έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τις χώρες αυτές θα ξέρει ότι είναι πολύ ε, ευαίσθητες ε, οι χώρες αυτές. Στη Λιβύη και η Λευκορωσία δεν χρειάζεται καν να αναφέρω γιατί, αλλά και το ίδιο ισχύει και για την Ιεμένη. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να συμφωνήσετε με τις τροπολογίες αυτές προκειμένου να ενισχύσουμε το Κοινοβούλιο και στο σημείο αυτό γιατί πρόκειται για μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, αξιοποιεί η ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Αουτάλα ζήτησε να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ήταν πολύ ανοιχτός. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και την εξετασή τους. Δεν θέλω να μιλήσω για τις τροπολογίες μου. Θέλω να πω απλά ότι θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία τα έχει ήδη συμπεριλάβει ο εισηγητής σε ό,τι αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα και την απόδοση ευθυνών, σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθυνών, συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας, οι διατάξεις για τον ανεκτό χαρακτήρα των εγγράφων ισχύουν και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρώ ότι είναι καλή η συμπερίληψη και της πτυχής της συνοχή, γιατί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δίδει δάνεια, εγγυήσει βάσει αρχών οι οποίες συνάγουν και με τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητή έδειξε ανοιχτό πνεύμα αναφορικά με τις τροπολογίες που πραγματεύονται διάφορες ε, συγκρούσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι πλέον συμπεριλαμβάνεται σωστά και αυτή η πτυχή σε ό,τι αφορά και τις ε, χώρες στόχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕΠ μπορούν να θεωρηθούν και ως ένα μέσο για την βελτίωση μεταξύ άλλων και της ε, διαχείρισης της διακυβέρνησης κάποιων τέτοιων χωρών στόχου. Θεωρώ ότι και η παροχή δανείων μπορεί να συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατάλογο των χωρών, έχω κάποιες αμφιβολίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε ό,τι αφορά τον ανεκτό χαρακτήρα, την ε, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Και θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, η λίστα αυτή, ο κατάλογος αυτός να διευρυνθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά την πτυχή της αλλαγής του κλίματος. Θεωρώ ότι είναι φυσικό, είναι αυτονόητο να ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μια στρατηγική για την αλλαγή του κλίματο. Μια στρατηγική η οποία θα συνάδει και με την γενικότερη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Μια νέα τροπολογία λοιπόν θα ήθελα να υποβάλω είναι η παριθμόν. είναι τμήμα της τροπολογίας 74, όπου ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καταρτήσει στρατηγική για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Μέχρι το 2012 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προτείνει μια στρατηγική η οποία θα συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους παγκόσμιους στόχους που τίθενται αναφορικά με τον κλάδο αυτό, με τον τομέα αυτό. Και θα ενισχύσει τα project τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2α. Αλλά... Καλώς, θα δώσω στο σκιώδη ηγητή, στον κύριο Νικόλα Χουντή το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίως σοβαρή δουλειά και με την ε, επεξεργασία των τροπολογιών. Θεωρώ σκόπιμο να επαναλάβω τις δύο βασικές μας ενστάσεις σε σχέση με την έκθεση – λέγοντας ότι και τροπολογίες που κατατέθηκαν στη συνέχεια και αφορούν τα δύο αυτά ζητήματα δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Η πρώτη μας παρατήρηση είναι η σύνδεση της δράσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τους εξωτερικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την ευκαιρία να σας πούμε ότι δεν συμφωνούμε με την εξωτερική πολιτική. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι λαθεμένη και η σύνδεση της δράσης της ΕΤΕΠ με αυτή την, ε, τον προσανατολισμό κατά τη γνώμη μας δεν είναι σωστό. Και το δεύτερο, η σύνδεση της ε, δράσης της ε, και η συμμετοχή στον προγραμματισμό ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με την ΕΤΕΠ και αυτό μας βάζει σε μεγάλες ανησυχίες. δεν θέλω να επαναλάβω τους, γιατί έχουμε πει τα επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει, όσες τροπολογίες ενισχύουν αυτές τις κατευθύνσεις δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Δεύτερο, στις αρχικές τροπολογίες φυσικά του εισηγητή είμαστε σύμφωνοι όσο αφορά την αύξηση των ανωτάτων ορίων χρηματοδότησης και το ότι πράγματι ε, προτείνει μέτρα ή εν πάση περιπτώσει ε, ε, βλέπει τον τρόπο αντιμετώπισης ούτω ώστε αυτοί οι εγγυήσει που δίνονται να εξασφαλίζουν ότι δεν θα έχουμε φοροδιαφυγή και δεν θα έχουμε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα. Τέλος, γιατί δεν θα ήθελα, είδα δεν υπάρχει ο χρόνος να αναφερθώ αναλυτικά στις άλλες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ε, σας είπα τα δύο κριτήρια με, τα οποία απορρίπτουμε παρόμοιες ε, παρεμφερείς τροπολογίες, όμως έχουν κατατεθεί και τροπολογίες που μας βρίσκουν σύμφωνους και αναφέρομαι στην κατηγορία γενικά ως κατηγορία τροπολογιών που έχουν να κάνουν πρώτον με την πρόθεση της διαφάνειας στον τρόπο της δράσης της ΕΤΕΠ, εκεί είμαστε σύμφωνοι, Δεύτερο, στη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Οι τροπολογίε αυτέ μα βρίσκουν σύμφωνος. Και τρίτο, τροπολογίε που αφορούν στην ύπαρξη κριτηρίων που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντο. Αυτέ τις τροπολογίε θα τι υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για να δώσει απαντήσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα λάβει χώρα αύριο, 5η 28 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου. Τα συμπεράσματα στον εισηγητή, τον συνάδελφο Πηγιού. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ τους τρεις συναδέλφους που πήραν το λόγο, Λάντσβορφ, Ουτάλα και τον κύριο Χουντή, που μίλησαν είδαμε ότι όσον αφορά τη διαφάνεια, τον έλεγχο, την αποτελεσματικότητα, προοδεύσαμε συνεργαζόμενοι. Όσον αφορά αυτό που η κυρία Χαουτάλα, τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο, δεν νομίζω ότι μα δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Όλε αυτέ οι απαιτήσει δεν είναι υπερβολικές. Ανησυχώ περισσότερο από αυτά που μας επανέλαβε και πολύ σωστά και με πειθό που συμμερίζομαι ο κύριος Λάμσντορφ. Πρέπει να βρούμε μια λύση κατά τη διάρκεια της μέρας, το επαναλαμβάνω αυτό, όντως ώστε ο κατάλογος των χωρών και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιμετωπίζουμε και η δυνατότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να ελέγχουν αυτές τις ευαίσθητες χώρες και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αυτές τις χώρες, να είναι κάτι ρεαλιστικό, λειτουργικό και ταυτόχρονα στεναρό. Θα επανέλθουμε του προβλήματος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους εκ νέου. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα που φέρνει αντιθέτους. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία πιστεύω. Θα πρέπει να βρούμε ίσως τη σύνταξη του κειμένου που θα προτείνεται να βρούμε τον τρόπο να το εκφράσουμε με τον σωστό τρόπο δεν λέω ότι είναι ευφυές να εξαιρέσουμε. ή Ίσως θέλουμε σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά τις χώρες αυτές. Είναι σωστή κατεύθυνση, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της μέρας και ελπίζω αύριο να έχουμε την καλύτερη δυνατή ψηφοφορία επί ενός κειμένου που ίσως φαίνεται για μερικού πάρα πολύ τεχνικό το κείμενο, αλλά όσον αφορά τις πολιτικές συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πεγιόν, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε στο επόμενο σημείο. Λοιπόν, ε, συνεργασία του πολιτικού και στρατιωτικού ταμεία. Ε, ο κύριος Χέλερ παρουσίασε το θέμα στις 27 Σεπτεμβρίου. 157 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Οι τροπολογίες, οι 11 τροπολογίες συμβαστικές που προτείνονται από τον εισηγητή ήδη συζητήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου. Οπότε θα πρέπει να περιοριστούμε στη σύνοψη των βασικών θεμάτων. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη το πρωί. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Έλλερ. Συνάδελφοι, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες ε, της Επιτροπής για την επικοτομητική εργασία ξεκινήσαμε με ένα εμπειρικό έγγραφο, όχι με ένα προσχέδιο για την ε, κατάσταση ως έχει, εμπειρικά σε ό,τι αφορά την στρατηγική συνεργασία και τα σχετικά μέσα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μαζί αναπτύξαμε το πώς, ε, την ιδέα για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί η θέση του Κοινοβουλίου στη συζήτηση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι μπορέσαμε να διατυπώσουμε να υποβάλουμε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες και να διαμορφώσουμε την ε, έκθεση με πολύ καλύτερο τρόπο. Να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση. Δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία όπου αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια πολιτικο-στρατιωτική προσέγγιση στις κρίσεις και ότι οι αμυγός πολιτικές ή στρατιωτικές ε, προσεγγίσεις μπορεί να είναι επαρκείς. Στην τροπολογία 3, τη συμβιβαστική τροπολογία 3, μιλάμε για τους ε, μη κρατικούς φορείς σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Τέταρτος συμβιβαστική για τη σχέση μεταξύ των πρώην ε, υπηρεσιών της Επιτροπής και των δομών της ΚΕΠΑ σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των μέσων που χρηματοδοτούνται από τα μέσα σταθερότητας και σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ EAS και τα ονογραφείων του, της ΚΕΠΑ. Αυτά είναι σημαντικά. Στις διαθεσμικές ε, διαδικασίες στην συμβαστική 4 αναφέρεται ότι δεν μιλάμε για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να βασιζόμαστε στην ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Συμβιβαστική 6 που τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ισορροπημένης ε, στρατιωτικής ε, πτυχής στο, και στην ΚΕΠΑ. Η συμβιβαστική 7 τονίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και ζητά να γεφυρωθούν οι δύο διαδικασίες ε, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας και αυτό υπό τους ε, στόχους ε, επικεφαλίδας. Στη συμβαστική εννέα είναι πολύ σημαντική γιατί τονίζει τις τροπολογίες που τονίζουν τον ε, ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Στην τροπολογία 11 τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης αυτονομίας σε ό,τι αφορά μεταξύ τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και νομίζω ότι επί της αρχής συμφωνήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη από πλευρά του Κοινοβουλίου να υπάρξει μια συνεκτική έκθεση, να μην κάνουμε αναφορά σε αφηρημένα πολιτικά θέματα, να διατυπώνουμε συγκεκριμένες θέσεις στις συζητήσεις για την εκ νέου διαμόρφωση των δομών πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας. Άρα, επί της αρχής βασιστήκαμε σε τρία θέματα. Βελτίωση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και νομίζω ότι εκεί καταφέραμε να επικεντρωθούμε σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η ανάπτυξη στρατιωτικών εικονοτήτων. Αναφέραμε θέματα αντιμετώπισης ε, κρίσεων ε, στελέχωσης, εκπαίδευσης, διεθνικής ε, συνεργασίας. Δεν μπορέσαμε να αποτεχτούμε τις ε, τροπολογίες που αρνούνταν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τέτοιο μηχανισμό, τέτοιες δομές. Νομίζω ότι αυτό θα μα δώσει μια άλλη δύναμη στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος ο κύριο Λούζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, επειδή χτε ε, εξέφρασα την θέση της ομάδας μου στην Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κρίσης και υπέβαλα σχετικές τροπολογίε. θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ μόνο μία στιγμή εξ ονόματος της ομάδας μου τίθεμαι κατά οποιοδήποτε μέτρο πολιτικο-στρατιωτικού. Με την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία γίνεται διάκριση μεταξύ, μάλλον δεν επιτρέπεται διάκριση μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτική σκελου. Απαιτούμε αμυγό πολιτική δύναμη, ειρηνική δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, ε, γιατί συχνά αναφέρεται ότι είναι απαραίτητα τέτοια μέτρα για τους ε, οργανώσεις βοήθειας. Και οι ενώσεις όμως βοήθειας ε, αναφέρουν ότι αυτά τα μέτρα τις εμποδίζουν, δεν τις βοηθούν. Αναφέρεται ότι πολλές φορές χρειάζονται τέτοια μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό. Αλλά κοιτώντα τι εφημερίδε, έχουν την εντύπωση ότι οι πολίτες θα πρέπει να προστατευτούν από το στρατιωτικό σκέλο. Δεν είναι η στρατιωτικό σκέλο που προστατεύει τους πολίτες. Αντίστροφα, θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα του πολιτικού σκελου. Όπως είπα και χτες, στην έκθεση αυτή δεν υπάρχει κανένα σημείο για το οποίο δεν μας βρίσκει έντονα αντίθετους και εξήγησα ποια σημεία με βρίσκουν αντίθετοι θα πρέπει, μάλλον οι τροπολογίες ε, κατευθύνονται προς την πλευρά της βελτίωσης, αλλά και πάλι θεωρούμε ότι το κείμενο και με τις τροπολογίες αυτές δεν θα ήταν επαρκές. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμφωνήσω με την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καλημέρα και σας ευχαριστώ. Όπως είπε και η συνάδελφος, θα συζητήσαμε τα θέματα αυτά και χτες. Θα ήθελαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποβολή της έκθεσης αυτής και για τα θέματα τα οποία εξηγήσατε και για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες τις οποίες αποστήλετε χθε το βράδυ. Με την τροπολογία 4, τη συμβιβαστική 4, πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε. Χαιρόμαστε που συμπεριληφθήσε για τα άλλα θέματα σε ό,τι αφορά την απαρίθμηση των διάφορων αποστολών και το τι υπάρχει, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν καλό για την ε, ε, για το ψήφισμα, θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε. Λοιπόν, χτες ανέφερα και το θέμα για την ε, Disaster Release Crisis Response. Νομίζω ότι και στην έκθεση Weber την οποία συζητούμε, πολλά θέματα ήταν κοινά και από τους δύο αρμόδιους ε, άκουσα ότι υπάρχει ένας τομέας αλληλοεπικάλυψης θα πρέπει όμως να είμαστε συνεπεί μεταξύ των δύο εκθέσεων. Δεν μπορούμε στην έκθεση Βέβρου να λέμε άλλα από την έκθεση αυτή. Θα πρέπει, γιατί ακριβώς επειδή γίνεται και παράλληλα αυτή η συζήτηση, θα πρέπει να αναρμονιστούν οι δύο εκθέσεις. Γιατί θα τις ψηφίσουμε άλλωστε και την ίδια μέρα. Να κάτσουμε να τα συζητήσουμε αυτά, να υπάρχει μια συνεκτική θέση του Κοινοβουλίου, να ψηφίσουμε κάτι συνεκτικό την Πέμπτη για την 84, την τροπολογία 84, το θέμα του προσωπικού από το κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Από μια περσινή έκθεση προκύπτει ότι το ποσοστό είναι 31,7%. Ίσως θα έπρεπε να διαγράψουμε το τι αποστολές. βρίσκονται σε καθεστώς ανοιχτού καθεστώτος. Αν κάποιες ε, αποστολές έχουν ε, πολύ περιορισμένο προσωπικό, ίσως θα χαιρόντουσαν μερικές χώρες να συμμετάσχουν, να αποστείλουν πιο πολλά μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να ε, απευθύνουμε τέτοιες εκκλήσεις για αποστολή ίσως πολιτικού προσωπικού. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προφορική τροπολογία, να πούμε ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ε, αξιοποίηση προσωπικού τηρωμένων των γεωγραφικών ε, ισορροπιών. Ανέφερα και κάποια στοιχεία χτες, όπως για παράδειγμα το θέμα της έρευνας άμυνας και της συμπερίληψής της στην έκθεση για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είμαστε κατά της, 30, της 131, η οποία αν περάσει θα καταψηφίσουμε ε, την έκθεση. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες ε, μάχης. Θεωρούμε ότι αρκεί να προστατεύσετε ο Πληθυσμό ο άμαχο. Το Κονγκό αποτελεί ένα καρό παράδειγμα όπου γίνονται βιασμοί, δολοφονίε παιδιών. Εκεί μπορούμε να συνδράμουμε δηλαδή. Αν θέλαμε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα battle groups θα ήταν καλύτερο τρόπο. Αν περάσουν δηλαδή και οι 107 και οι 108 και πάλι μάλλον θα καταψηφίσουμε την έκθεση. Και τώρα ο σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Μαυρονικόλας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφέρω ότι με, το, με την αναφορά αυτή για πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και για δυνατότητες πολιτικοστρατιωτικές αγγίζεται ένα θέμα για πρώτη φορά Άρα και το κείμενο αυτό θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από την ε, προσπάθεια η οποία γίνεται για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα όσο το δυνατό πιο σφαιρικά, πιο αντικειμενικά, αλλά να δοθούν και διάφορες προτάσεις οι οποίες να είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη πολιτικών και στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων συνεργασίας. Θα ήθελα από την πλευρά μου να τονίσω ότι το κείμενο κατά τη δική μας άποψη είναι πολύ ικανοποιητικό, όπως επίσης να εκφράσω και την ευαρέσκειά μου για τη στάση του Κρίστιαν σε όλες τις προσπάθειες για να δομηθεί ένα κείμενο το οποίο να είναι αντικειμενικά αποδεκτό από όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές ομάδες. Είναι ένα κείμενο το οποίο αποδέχεται τις ευαισθησίες οι οποίες υπάρχουν και πολλά, πολλές από τις τροποποιήσεις που έχουμε προτείνει ως σοσιαλιστές έχουν αποσυρθεί μέσα από την δυνατότητα ε, ε της σύνταξης αυτών των compromise που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το κείμενο αυτό αγγίζει ε, και διαχωρίζει και το πολιτικό και το στρατιωτικό τμήμα δίνοντας ακριβώς μια δυνατότητα κοινή δράσης, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ιεραρχίας, δίνει προτάσεις για το πώς μπορούν να επεκταθούν ε, οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά και πώς μπορούν να συμπληρωθούν οι αναγκαίες ε, εγκαταστάσεις για να δοθεί η δυνατότητα κοινών αποστολών όπως επίσης αγγίζει θέματα τα οποία αφορούν ε, το EAS, e δηλαδή την εξωτερική πολιτική, τη σύνδεση του θέματος αυτού με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών. Είναι ένα ικανοποιητικό κείμενο. Νομίζω ότι οι δικέ μας αλλαγές οι οποίες ζητούνται πλέον είναι ελάχιστες και πιστεύω ότι η σοσιαλιστική ομάδα θα υπεψηφίσει στην αυριανή ψηφοφορία έναν κείμενο αντιπροσωπευτικών και αντικειμενικά, αντικειμενικών δυνατοτήτων για να βάλει για πρώτη φορά το θέμα κάτω ε, για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Αρλάκη, αλλά παρόλα. Αρλάκη, ο κύριος Αρλάκη. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις έχω. Δεν γνωρίζω πολύ καλά το πώς διαμορφώθηκε η έκθεση. Διάβασα το κείμενο και κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Και ελπίζω ότι οι τροπολογίες θα βελτιώσουν το κείμενο. Θα το καταστήσουν πλέον εύληπτο, ευνόητο ακριβέστερο. Διότι διάβασα το κείμενο και δεν κατάλαβα τι είναι αυτή ε, η πολιτικοστατιωτική ικανότητα και η πολιτικοστατιωτική συνεργασία. Ξέρω λίγο τα πράγματα, τα θέματα αυτά και το πρόβλημα είναι δεν περιέχονται στοιχεία. Ούτε ορισμός της δομής, ούτε συνέπειες για τον προπολογισμό. Πόσο κοστίζει αυτή η δομή, πόσο προσωπικό θα απασχολείται και ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός. Και όσον αφορά τις άλλες υπηρεσίες, τους άλλους φορείς, αναφέρεται το ΝΑΤΟ και πρόσκληση, έκκληση στο ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί όσον αφορά το πολιτικό δυναμικό, κάτι κατανοητό σαν αρχή, Είδα κάποια άλλη αναφορά για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΟΗΕ. Πολύ αοριστό το κείμενο. Δεν λέει τι πρέπει να κάνει αυτή η πολιτικοστατιωτική ικανότητα που δημιουργείται όσον αφορά την ε, ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς σε κάποιον τι θέλουμε να κάνουμε, τι πρόκειται να κάνουμε στην πραγματικότητα. Ελπίζω ότι οι τροπολογίες θα κάνουν πιο κατανοητό το κείμενο, πιο συγκεκριμένο. Καταρχήν, συμφωνώ με την ιδέα και ελπίζω η ιδέα να γίνει πιο συγκεκριμένη με μια πιο καλή διατύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αλάκη. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι από τις πιο σοβαρές προκλήσεις. Πώς θα συνδυάσουμε την πολιτική με τη στρατιωτική συνεργασία. Και νομίζω ότι ο κύριος Σέλερ απάντησε με πολύ ανοιχτό, κατανοητό και εξαιρετικό τρόπο. Εγώ συμφωνώ με τις συμβαστικές τροπολογίες. Το θέμα είναι πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η συνεργασία και πώς θα βελτιωθεί και ο συντονισμός. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια των πολιτικών ικανοτήτων. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της τροπολογίας 47 που ζητά ενίσχυση των άρθρων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την αμοιβαία αρρωγή και την επίδειξη αλληλεγγύης. Είναι σημαντική και η διοργανική συνεργασία μεταξύ της νέας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και των λοιπόν θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια έγκαιρης αντίδρασης και συντονισμού από την αρχή, από τις πρώτες ώρες δηλαδή οποιασδήποτε εκτάκτο ανάγκης που παρατηρηθεί. Εγώ είμαι υπέρ του γράφου και εύχομαι καλή τύχη στον εισηγητή τον κύριο Έλλερ. Ε, εισηγητής, κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Θεωρώ ότι ως κοινοβούλιο το έργο μας είναι κατά την διατύπωση των ε, δομών αυτών να συζητήσουμε τέτοια θέματα γιατί βρισκόμαστε, κατά τη διάρκεια, βρισκόμαστε στη διάρκεια της ε, διαμόρφωσης τους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ενιαία θέση. Να πούμε στην κυρία Λέζε ότι τη γενική κριτική για τις στρατιωτικές δυνάμεις με ενθάρρυνε να προχωρήσω προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν με αποθάρρυνε. Δύο πτυχέ είναι σημαντικές για τα battle groups. Δεν ισχύει αυτό που είπε η κυρία Μπράτνερ. Δεν επιδιώξαμε να χρησιμοποιούνται για προστασία από καταστροφές. Επιδιώξαμε τα battle groups να προσαρμόζονται, να έχουν δυνατότητα προσαρμογής. Αν μία αποστολή είναι για παράδειγμα, στρατιωτική φύση και αλλάξει η φύση τη γίνει πολιτική. Στα πλαίσια μιας πολιτικής, για παράδειγμα, αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο και ένα στρατιωτικό σκέλος. Το θέμα δεν είναι τα battle groups να χρησιμοποιούνται για ε, πολιτικές ε, ε αποστολές. Επίσης είπατε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Κοιτώντα τι εταιρολογικέ σκέψει τη έκθεση, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνδιάσκεψη, διατυπώναμε νέου στόχου. Συζητήσαμε εκτεταμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε τρει μεγάλε αποστολέ με 10.000 άτομα σε τρία έτη. Αυτό όμως που δεν κάναμε επί 10 χρόνια είναι να συζητήσουμε το πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Και από την άποψη αυτή θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο κλήθηκε να πει με σαφήνεια ότι κοιτάξτε υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των στόχων που έχουν διατυπωθεί και της επιχειρησιακής πραγματικότητας. Βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που θα πρέπει πλέον να διαμορφωθούν ε, οι δομές. Τέρμα πια στις πολιτικές ε, εκκλήσεις. Να δούμε ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις πρακτικά για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους που διατυπώθηκαν και θεωρώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η έκθεση αυτή. Ασχολείται με πρακτικά ζητήματα και μάλιστα με την υποστήριξη όλων των ομάδων της, ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο, πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό η συζήτηση επί του κύματος του ψηφίσματος δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα καλύτερη στιγμή. Τους τελευταίους μήνες έγιναν σημαντικά πράγματα για τη Σερβία και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σερβίας. Ξεκίνησε η διαδικασία επικύρωση της Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης. Υπήρξε ψήφισμα συμβιβαστικό όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο και είχε θετική έκβαση στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και υπήρχαν εντάσεις στο Βελιγράδι πρόσφατα και στις 25 Οκτωβρίου αποφάσισε το Συμβούλιο να στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Σερβίας, την επίσημη αίτηση ένταξης. Η γνωμοδότηση λοιπόν του Κοινοβουλίου όσον αφορά τι εξελίξει στη χώρα έχουν μεγάλη σημασία θα δώσω το λόγο αμέσως στο συνάδελφο τον κύριο Κάτσιν, ο οποίος είναι ο εισηγητής, για να παρουσιάσει την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την, για την απόφαση του Συμβουλίου της Δευτέρας που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφέρει γνώμη σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα τη Σερβία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το μήνυμα που στέλνουμε στο Βελιγράδι και ε, ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο τη ενταξιακή διαδικασία τη Σερβία στην Ευρώπη. Και όσο εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, έκθεσή τη για το Βελιγράδι θα μπορέσει να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα επιτεύγματα της Σερβίας αλλά και την πρόοδο που θα κληθεί να πραγματοποιήσει στο μέλλον. Δημιουργήθηκε μεγάλη αισιοδοξία στο Βελιγράδι και νομίζω ότι θα δοθεί και το έναυσμα για θετικές εξελίξεις. Η έκθεση που εξετάζουμε σήμερα παρακολουθεί αυτές τις θετικές εξελίξεις Φυσικά εκδηλώνουμε πνεύμα συνεργασία, αλλά επισημαίνουμε και τα προβλήματα που θα πρέπει να υπερκεραστούν. Καταρχήν, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία και το Κωσυφοπαίδιο. Η συνεργασία τη Σερβία με το δικαστήριο αυτό ήταν σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση τη πρόοδου τη χώρα αυτή προ την διαδικασία τη ένταξη. Ο Κόραν Χάτζη και ο Βλάτκο Τάντιτς. Μερικοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσει στο Βελιγράδι για να σημειώσει ακόμη πιο εντυπωσιακά βήματα πρόοδου. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να στείλει το έγγραφό της στο Συμβούλιο και να επισημάνει στη Σερβία ότι αν δεν κλείσει αυτό το κεφάλαιο δεν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να δώσει θετική γνωμοδότηση για την υποψηφιότητα της Σερβίας αν δεν κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την, έκθεση, την ε, Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μετά το ψήφισμά μας. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται να γίνει αν δεν συνεργαστεί προηγουμένως η Σερβία με το δικαστήριο της Χάγης και αν δεν εκδώσει τους Χάτζης και Κάρατζης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας. Σε ό,τι αφορά το Κωσυφοπαίδιο, πέραν της συνεργασίας με το Δικαστήριο της Χάγης, η Σερβία θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τις γειτονικές της χώρες. Γιατί είναι αρκετά ταραχώδεις οι σχέσεις που έχει η χώρα αυτή με τις γειτονικέ της χώρες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μία πρόοδος. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έγκριση του ψηφίσματος για τη Σερεμπρένιτσα στη Σερβική Βουλή. Επίσης το θέμα της ανακήρυξης ανεξαρτησίας του Κουσυφοπεδίου ήταν από τα σημαντικά προσκόμματα ε, για τις ε, καλές σχέσεις της Σερβίας με τις γειτονικές σχέσεις. Πάντως ε, επικροτούμε την προθυμία της Σερβίας να έχει διάλογο με την Πρίστινα. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συμμετέχουν στο διάλογο για να γίνει καρποφόρος και επικοδομητικός. Και προσβλέπουμε στην άμεση έναρξη αυτού του διαλόγου με συμβιβαστικό πνεύμα από τις δύο πλευρές προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενταξιακές τους φιλοδοξίες. Είναι σημαντικό και το θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης Σερβία και την εξασφάλιση του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει όλες τις ε, μεταρρυθμίσεις της Σερβίας, αν και στο πρόβλημα της δικαστικής μεταρρύθμισης ε, η κατάσταση χωλαίνει, όπως επισήμαναν οι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τους 850 δικαστές που διορίστηκαν ε, στις εκλογές, μόνο οι μισοί έχουν λάβει μια απάντηση για τις αιτιάσεις τους. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δυστυχώς έχουν απομείνει και πολλές εκκρεμότητες στο θέμα αυτό. Η δικαστική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πάταξη της διαφθοράς είναι ένα θέμα φυσικά άμεσα συνδεδεμένο με το, την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Και σίγουρα η ο Οργανισμός για την Πάταξη Διαφθοράς θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος από τις υπόλοιπες κρατικές δομές. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή των περιουσιών, και εκεί σημειώθηκε πρόοδος, αλλά όχι αρκετή. Ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με βάση τους α, ε, δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, η Σερβία πέρασε από τη θέση 62 στη θέση 85 και δυστυχώς ε, ο σκαδαλοθερικός τύπος ε, είναι αυτός περισσότερο ανθεί στην Σερβία και έχουμε και δυστυχώς απειλές κατά των δημοσιογράφων. Είναι πολύ σημαντικό και το θέμα των απαντήσεων που θα πρέπει να λάβουμε στις ερωτήσεις που στείλαμε, γιατί δημιουργούνται δυστυχώς εμπόδια στην ομαλή συνεργασία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Ελπίζω ότι η Σερβία θα ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες γιατί βρίσκεται πραγματικά σε ένα ιστορικό ταξίδι για την ενδεχόμενη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όσο πιο σαφείς γίνεται, να δώσουμε την ε, ισχυρή μας υποστήριξη προς τις σερβικές προσπάθειες, αλλά να τονίσουμε και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η σερβική ηγεσία. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του ψηφίσματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου και τη γραμματεία της ΑΦΕΤ για τη βοήθεια που μου έδωσαν κατά την κατάρτιση του ψηφίσματος. Και επίσης ε, να ευχαριστήσω τη Μίλτσα Ντέλεβιτς για την ε, πολύ επικοδομητική προσέγγιση που είχε στις ε, συνομιλίες μας. Σας ευχαριστώ και είμαι ανοιχτός προς τη συζήτηση και περιμένω τις ερωτήσεις σας για να δώσω απαντήσεις. Ευχαριστώ. Η παρεμβάση των σκιωδών εισηγητών. Κύριε Σλέφλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, πίσω. Ευχαριστώ τον κύριο Κάτσεν. Η έκθεση είναι πολύ καλή, διεξοδικότατη, καλύπτει όλα τα σημαντικά ζητήματα. Η Σερβία άρχισε να κινείται προς την Ευρώπη. Προφανώς αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Είναι θεμητό να πούμε ότι η διαδικασία είναι αργή και δεν θα γίνει εν μία νυχτή αλλαγή. Ε, είναι σημαντικό οι σερβικές αρχές και η κοινωνία της Σερβίας να κατανοήσουν ότι χρειάζεται χρόνος. Όμως είναι κάτι το οποίο θα συμβεί. Συμφωνώ απολύτως ότι η πλήρης ε, συνεργασία με το Διεθνές ε, Δικαστήριο αποδοχή του κοσυφοπεδίου ως μια πραγματική οντότητα είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη όμως θα έλεγα ότι δεν αρκούν αυτές καθεαυτές. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που εκκρεμούν. Σχεδόν όλα περιέχονται στην έκθεση του κυρίου Κατσίν πριν να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης η Σερβία. Αυτό που δεν βρήκα στην έκθεση είναι ένας δύσκολος τομέας. Ότι εξακολουθούν να επικρατούν οι μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα κρυμμένο κάτω στη Σερβία αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί πριν γίνει πλήρης δημοκρατία της Σερβίας, διότι στρεβλώνεται έτσι η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και διάφορες μορφές πολιτικής παρέμβασης που ανέφερε ο κ. Κάτσιν στην εισαγωγή του εν μέρη οφείλονται σε αυτό το γεγονός. Η διαφθορά ε, είναι σημαντικό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει μακρά ιστορία του προβλήματος, σε κάποιο βαθμό ήδη υπήρχε κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περίοδου και μετά επιδεινώθηκε σαν αποτέλεσμα μέρη του του παγκοσμίου μποϊκοτάζ κατά της Σερβίας αρχές της δεκαετίας του 90, αυτό επιδίνωσε τη διαφθορά και είναι πολύ δύσκολο να εκριζωθεί. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες μαφίες, την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα που ανέφερε ο κ. Κατσίν, Πέραν αυτού θα προσέθετα ότι χρειάζεται πολύ αυστηρότερος ε, διαχωρισμός εξουσιών από ό,τι υπάρχει τώρα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Οι ε, διάφοροι θεσμοί, ε, το κύρος των θεσμών, αυτό είναι ένα πρόβλημα σε όλες τις πρώην κομμουνιστικές χώρες, είναι το θέμα του κράτους δικαίου το κύρος των θεσμών παραμένει χαμηλό. Πολλοί θέλουν να χρησιμοποιούν γνωστούς διασυνδέσεις σε επαφές με το κράτος παρά να βασιστούν στις επίσημες διαδικασίες μέχρι ότου διορθωθεί αυτό, μέχρι ότου αποκατασταθεί ισορροπία. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για μια λειτουργούσα δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κάτσιν. Νομίζω ότι η Σερβία έχει πολύ κεντρική εξουσία και η αποκέντρωση της εξουσίας είναι κάτι σημαντικό θα ανέφερε όπως και εκείνο το θέμα της Βοηβοδίνας με την ε, πολυπολιτισμική της ε, φύση. Αναγνώριση αυτού είναι αναγκαία προϋπόθεση για να επικρατήσει η δημοκρατία στη Σερβία που όλοι θα επιθυμούσαμε. Τώρα, διόρθωση των σχέσεων με τους γείτονες. Αυτό σημαίνει επίσης να συμφιλειωθεί με το παρελθόν, όχι το πολύ πρόσφατο, την τελευταία 20 αλλά από όταν ε, έπεσε η κομμουνιστική εξουσία. Φρικτά πράγματα συνέβησαν το 44-45, εν μέρη αποκαλύφθηκαν, η Σερβία το έχει αντιμετωπίσει εν μέρη, αλλά μέχρι ότου η σερβική κοινωνία καταλάβει ότι έχει αρκετά δυσάρεστη ιστορία πίσω της, δεν θα μπορέσει να αναγνωρίσει τον εαυτό της και την πραγματική της υπόσταση και το απολευθερωμένο καθεστώ των θεωρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και θα ήταν άκρο λυπηρό αν υπονομευθεί κατά κάποιο τρόπο. Τέλο, για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τον κύριο Κάτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή έκθεση και ευχαριστώ όλου όσου συνεργάστηκαν μαζί του. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά, σκιώδη εισηγήτρια για το κομμάτι σου. Uh, like congratulate... Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή καταρχάς τον κύριο Κάτσιν για την ε, πλήρη έκθεσή του για τη Σερβία και όπως ήδη είπατε κύριε Πρόεδρε η πρόταση ψηφίσματος κατατίθεται σε πολύ σωστή χρονική στιγμή, δύο μέρες μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που πήρε απόφαση να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει την νομοδότησή της και μερικές μέρες πριν από την έκθεση Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε διάφορου τομεί και τι προσπάθειε που έχουν καταβληθεί από τη σερβική κυβέρνηση, ούτω ώστε να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει τη στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού τη χώρα, κάτι που η πολιτική μα ομάδα, οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε υποστηρίζουμε πλήρω. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι η Σερβία είναι σε ένα σταυροδρόμι η θέση μας και ενώ η θέση της Ευρώπης θα καθορίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει αυτή η χώρα, θα καθορίσει τη σταθερότητα και το μέλλον της Σερβίας και συνεπώς και της περιοχής των Βαλκανίων εν γέννη. Η Σερβία χρειάζεται την Ευρώπη και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τα ευρωπαϊκά δυτικά Βαλκάνια χωρίς τη Σερβία. Βεβαίως και συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή, είναι στα χέρια της σερβικής κυβερνήσεως και του σερβικού λαού η πρόοδος και αντιμετώπιση των επικειμένων προκλήσεων. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι η Σερβία του 2010 δεν έχει καμία σχέση με τη Σερβία του 2000. Η χώρα έχει μια πραγματικά δημοκρατική κυβέρνηση που κινείται προς ευρωπαϊκές προοπτικές και θέλει να γυρίσει σελίδα. Και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η Σερβία έδειξε πρακτικά την αποφασιστικότητά της να κινηθεί προς την Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω τη μονομερή εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας, ε, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της Σερβίας Σερμπενίτσα, το αίτημα για ένταξη στις 27 ε, ε, Νοεμβρίου του 2009 και επίσης και η συμφωνία για άμεσο διάλογο με το Κωσυφοπέδιο από την αιγίδα της Ευρώπης. Όμως η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δύο εμπόδια, το Κωσυφοπέδιο από τη μία πλευρά και το διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο από την άλλη η επίλυση του προβλήματος του κοσυφοπεδίου δεν είναι προπετούμενο όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο, όμως ξέρουμε ότι η εξέλιξη όσον αφορά το κοσυφοπεδίο θα είναι κρίσιμου σημασία για τις προπτικές της Ευρωπαϊκής Σερβίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, το συμβαστικό ψήφισμα του ΟΗΕ είναι ένα σωστό ε, βήμα για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και των αρχών ε, του Κωσυφοπεδίου. Ο συγητής σοφά διάλεξε ναι, να μην αναφερθεί εκτενώς στο θέμα του Κωσυφοπεδίου. Η πολιτική μου ομάδα ευθύς εξ αρχή είχε υποστηρίξει τον άμεσο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, κάτι που σίγουρα θα επηρεάσει θετικά ε, τις ευρωπαϊκές προοπτικές της δημοκρατίας της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Δοθήσει στις δύσκολης πολιτικής καταστάσεως στην Πριστίνα θα πρέπει να προσθέσουμε στην παράγραφο 4 τι περιμένουμε από το διάλογο. Ίσως να αναφέρουμε μια σταδιακή προσέγγιση η οποία θα επιτρέψει την έναρξη του διαλόγου του ταχύτερο δυνατόν, ένας διάλογος που πρέπει να ξεκινήσει από τις πλέον τεχνικές πτυχές και να συνεχίσει με τα πιο δύσκολα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η ειδική αναφορά χρειάζεται στη σημασία που έχει για τη συνεργασία της Σερβίας με τη Γιούλεξ, που είναι κάτι που κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την αναφορά του στο, στην παράγραφο 5, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι για ε, ειρηνική συνεργασία, πολιτική σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή και όλα αυτά περνάνε από αναγνώριση των παλαιών εγκλημάτων, αναγνώριση των εγκλημάτων πολέμου και συμφιλίωση. Όλοι συμφωνούμε ότι η πλήρη συνεργασία και η σύλληψη των ελαχίστων φυγοδίκων είναι κάτι που έχει προτεραιότητα. Τι σημαίνει η καλή συνεργασία. Μπορούμε να υπονοήσουμε ότι οι σερβικές αρχές δεν συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι ένα θέμα ερμηνείας και η ερμηνεία ανήκει στο ίδιο το ποινικό δικαστήριο. Η σύλληψη βεβαίω είναι η τελική απόδειξη της συνεργασίας, αλλά η πλήρη συνεργασία δεν ταυτίζεται με τη σύλληψη. Εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της ενταξιακής της Σερβίας μπορούμε να αξιολογήσουμε, και αυτό αναφέρεται και στα συμπεράσματα άλλωστε, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Δευτέρας, κατά πόσο υπάρχει αυτή η πλήρη συνεργασία ή όχι. Το τελευταίο θέμα που έχω να θίξω αφορά την αναφορά του εισηγητού στην ίδια παράγραφο, στην ανάγκη που υπάρχει να επαναξεταστεί όλη η στρατηγική για να εντοπιστούν οι φυγάδες. Ε, αυτά είναι αόριστα. Ποια είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική που θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Υπάρχει τέτοια στρατηγική. Ίσως θα ήταν πιο παραγωγικό να αναφερθούμε σε ερευνητικέ μεθόδους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 49 της προηγούμενης εκθέσεως και καλείται εκεί η Σερβία να αυξήσει τη συνεργασία της και να υιοθετήσει πολυσχηδή προσέγγιση για την σύλληψη των φυγοδίκων. Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συνεργασίας πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι η πρόσφατη ανακάλυψη του ημερολογίου του προσωπικού του Μλάντιτς με χιλιάδες φελίδες που δίνει πολύτιμες πληροφορίες στη δικαιοσύνη για δραστηριότητε του φυγοδίκου και του πολέμου. Θα ήθελα τώρα να στραφώ σε άλλο σημαντικό σημείο που είναι σημαντικό για μας. Η περιφερειακή συνεργασία είναι ακρογωνίω λήθο για την πολιτική μα στα Δυτικά Βαλκάνια και θα πρέπει να προσθέσουμε μια αναφορά και ενθαρρύνουμε τη Σερβία να δραματίσει επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή και να εργαστεί ρεαλιστικά σε όλα στα περιφερειακά φόρα. Στην παράγραφο 3 για την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επιστολή της Επιτρόπου Μάλστρομ και να δώσουμε προσοχή στα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα και πιστεύω ότι στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να προσθέσουμε επαφές λαού με λαό για να αναφέρουμε στη διευκόλυνση ε, ανταλλαγών στο πανεπιστημιακό επίπεδο θα ήθελα να προτείνω να αναπτυχθεί περαιτέρω παράγραφο 11 μέσω προσθήκη που επενεί την πρόοδο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο με δίτερη ερμηνεία στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Στην παράγραφο 10 που αναφέρεται στην συνεργασία με τονικέ χώρε και μεταρρύθμιση του αστυνομικού τομέα, θα πρέπει να σημειώσουμε τη σύμφωνη, πρόσφατη συμφωνία με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που έχει σημαντική συμβολική αξία και να προσθέσουμε ότι η Σερβία μέχρι τώρα έχει υπογράψει συμφωνίε συνεργασίας με 18 ευρωπαϊκές χώρες. Πέραν αυτού, ας μην λησμονούμε ότι η Σερβία από το 2007 έχει δημιουργήσει το γραφείο του Διαμεσολαβητή, ένα νέο θεσμό προθυμένης δημοκρατίας με πολύ θετικό ιστορικό παρά τις ε, δυσκολίες. Τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά την αποκέντρωση και το πρόγραμμα αποκεντρώσης της Σερβίας που αναφέρεται στην παράγραφο 14. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή για τη χώρα και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις στη Βοηβοδίνα. Θα προσέθετα μια τροπολογία σε μια προσπάθεια πιο εξισορροπημένης προσεγγίσεως. Να συγχαρώ εκ νέου του, τον κύριο Κάτσιν για την έκθεσή του και να κάνω και μια πρόταση. Η έκθεση της χώρας, για τη χώρα θα δημοσιοποιηθεί. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 8 Νοεμβρίου. Θα μπορούσε να παραταθεί λοιπόν η προθεσμία της τροπολογίας που είναι 10 Νοεμβρίου για να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη αυτή την έκθεση. Αυτά και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Υπάρχει μακροσκελής κατάλογος αγοριτών και για να δώσω στον καθένα τη δυνατότητα να μιλήσει θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο στα τρία λεπτά για τον καθένα από, που θα πάρει, από εκεί θα πάρουν το λόγο, λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τι 12.30 τι εργασίε μα. Μπραντνερ, κυρία Μπραντνερ. Και παρακαλώ να τηρήσει το τρίλεπτο. Sorry, thank you. Um, we really, we spoken σας ευχαριστώ. Το ζητήσαμε και στην ομάδα εργασίας ε, το σχέδιο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό το κείμενο και βρίσκει σωστή ισορροπία. Θα ήθελα να θέσω κάποια σημεία. Η συναδελφό θα τονίσει και κάποια άλλα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά θεωρώ ότι συμφωνώ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος με το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να συμβεί αυτό, είναι στο βήμα, αλλά θα πρέπει παράλληλα να αφαιρεθούν σιγά σιγά οι δομές στο κουσικοπαίδιο του Σερβικές. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Μιλώντας για το κοσυφοπέδιο, να μην ξεχνάμε το βοσνιακό κράτος και την τάσμευση που υπάρχει για ένα ισχυρό και ενωμένο τέτοιο κράτος. Και εδώ θα πρέπει να είναι έντονη η διατύπωση. Και φυσικά ένα σημείο που ανησυχεί όλες τις χώρες ε, που είναι σε πορεία ένταξης είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού. Και όπως είπα, καλωσορίζουμε την ε, έγκριση της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στο Σερβικό Κοινοβούλιο και καλό να ολοκληρωθούν γρήγορα μεταρρυθμίσεις. Και τώρα να αφήσω το λόγο στην συνάδελφο Λίζε. Η κυρία Κούγκαν, που είναι της αντιπροσωπή την Ατελική Ευρώπη. Ο κύριος Κούγκαν, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι πολύ καλό και αγγίζει όλα τα σχετικά θέματα για τη Σερβία. Δέκα χρόνια μετά την εποχή του Μιλόσεβιτς, η Σερβία κάνει σημαντικά βήματα προ την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε γενικέ γραμμέ. Η Σερβία σημείωσε καλή πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Δύο, προγραμ, δύο παραδείγματα, συμφωνία σταθερότητα και η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση ενοποίηση να παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Σερβίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση αυτή και μια σημαντική θετική εξέλιξη είναι ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κάλασε να προετοιμαστεί μια γνωμοδότηση για τη Σερβία. Είναι θετικό αυτό, όχι μόνο για τη Σερβία, αλλά για όλη την περιοχή. Το τονίζω αυτό. Το συμπέρασμα του... Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αναφέρουν τον επικοδομητικό διάλογο και αναφέρουν ως προϋπόθεση την πλήρη ε, συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συνεκβανών, κοντίτσιο συνεκβανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, θα πρέπει να τονίσει τα σημεία αυτά και στο ψήφισμα. Πριν από κάποιες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκέφθηκε το Βελιγράδι και συζήτησε θέματα τα οποία σχετίζονταν με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Σερβία. Νομίζω ότι κάποια τα θέματα αυτά θα πρέπει να αναφερθούν και να εξεταστούν στην έκθεση. Καταρχάς, η περιφερειακή συνεργασία είναι σημαντικό σημείο που δείχνει την ικανότητα των χωρών να συνεργάζονται είτε σε δεμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο με τους γειτονές τους. Εν γέννη, η Σερβία μπορεί να επενεθεί για την προσέγγιση της αυτή. Το επίσης παραμένει το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας με το κοσυφοπαίδιο. Ένα άλλο θέμα είναι οι καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες της, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δύο θέματα μας απασχολούμε. Ο αυξανόμενος αριθμός ε, προσφύγων από την ε, Σερβία ετούντων άσυλο που δυσκολεύει το θέμα της που δυσκολεύουν τα πράγματα για τις θεωρήσεις για την Αλβανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ένα άλλο θέμα είναι ο εξτρεμισμός και οι ακραίες ομάδες στη Σερβία. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι ένα πρόβλημα χτεσινό αλλά ένα θέμα το οποίο είτε αφέθηκε στην τύχη του, είτε και έγινε κατάχρηση αυτού για πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, θα πρέπει να πάρει ένα τέλος, όσο και αν είναι δύσκολο να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Κάτσιν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος, ο κ. Ντανζόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γελκο Κάτσιν για την έκθεσή του που είναι πολύ εύστοχη, πολύ ισορροπημένη και προβάλλει και τις αναφυσβήτητες επιτυχίες της Σερβίας και της ε, κυβέρνησής της ε, στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένταξη και χαιρετίζουμε φυσικά, επικροτούμε αυτή την πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα δακτυλοδεικνύουμε και τις ελλείψεις και την πρόοδο που θα πρέπει να σημειώσει η χώρα αυτή στο μέλλον. Είναι πολλές οι επιτυχίες της Σερβίας, αλλά μερικές φορές ε, επαναπάβεται στις δάφνες της και χαλαρώνει την προσπάθεια. Είχαμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων, είχαμε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που ήταν σημαντική επιτυχία ε, για κοινή θέση Σερβίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κωσυφοπαίδιο. Επίσης έχουμε την εντολή του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ετοιμάσει την γνωμοδότησή της για την ένταξη της Σερβίας. Όλα αυτά είναι Εντυπωσιακέ πρόοδοι χάρη στην επιμονή και την αποφασιστικότητα τη σερβική κυβέρνηση. Αλλά δεν θα πρέπει να χαλαρώσει την προσπάθεια η σερβική κυβέρνηση. Θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα τι πιθανολογίες για, τη, για την ημερομηνία ένταξης. Ούτε η Σερβία θα πρέπει να δώσει τον πειρασμό να χαθεί σε αυτές τις οικοδολογίες. Επίσης θα πρέπει να ξεχνούμε και το θέμα της ανάγκης πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουκοσλαβία. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό και Νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε, να συμφιλιώσουμε μια τέτοια προϋπόθεση. Έχουμε την 10η επέτειο από την πτώση του Μιλόσεβιτς, έχουμε την 15η επέτειο από τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα. Είναι απαράδεκτο να εξακολουθεί να είναι ελεύθερος ακόμη ο Μπλάντης. Θα πρέπει να επιμείνουμε στη σύλληψη των εγκληματιών πολέμου και ταυτόχρονα να δείξουμε κατανόηση για την πρόοδο που έχει ακόμη να επιτελέσει η Σερβία. Κάθε μέρα ακούμε αποκαλύψεις για το τι δεν έγινε μεταξύ 2004 και 2008 από την προηγούμενη κυβέρνηση και χαιρετίζουμε το, τον ειδικό εισαγγελέα για τα εγκλήματα πολέμου πραγματικά με πολύ κουράγιο και θάρρος επιτελεί το έργο του. Πολλές ελλείψεις λοιπόν και παραλήψεις το 2004 με 2008. Θα πρέπει λοιπόν να επενέσουμε τη σερβική κυβέρνηση που θα πρέπει να συνεχίσει και το παιδαγωγικό της έργο γιατί η σύλληψη του Μλάντιτς δεν είναι τεχνικό ζήτημα ή πολιτικό μόνο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απόλυτη ανάγκη, ζωτική ανάγκη και για τη σερβική κοινωνία εξαιτία τη ε, έξαρση κάποιων ριζοσπαστικών φαινομένων που επισήμανε ο κύριο Σέπφλιν σε κάποιε κρατικέ δομέ. Ευχαριστώ. Τάλερ είναι το επόμενό μου, κύριο Τάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με το σχέδιο, με την πρόταση ψηφίσματος του κυρίου Κατσίν. Αυτό το κείμενο αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο τη Δευτέρα είναι θετική και από την εξή άποψη. Όταν η Σερβία απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που απεστάλλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα διλήμματά της. Πρόσφατα η Σερβία έχει δείξει ένα νέο πρόσωπο όσον αφορά κάποια θέματα, κυρίως όσον αφορά το ψήφισμα στον ΟΗΕ, όπου χρησιμοποιώντας ευφυή διπλωματία πρόεδρος Τάντιτς, 27 κράτη-μέλη και η Σερβία πέρασαν ένα συμβαστικό ψήφισμα. Και θα πρέπει να συγχαρούμε και την ύπατη εκπρόσωπο εδώ. Θα πρέπει αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να μην δεχθούμε καμία δικαιολογία όσον αφορά τις εκλογές και διάφορα άλλα ζητήματα, κυρίως αν η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο δεν θέλουν να σπαταλήσουν άλλη μια δεκαετία μέχρι ότου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους και μέχρι ότου να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δράσουμε τώρα. Μία σύσταση έχω εγώ Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο το Κωσυφοπαίδιο και η Σερβία να αντιμετωπίσουν τις σχέσεις τους στο ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και στο Κωσυφοπαίδιο και στη Σερβία. Θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο. Δυστυχώς υπάρχει και μια σκοτεινή όψη της Σερβίας. Αυτή συμπεριλαμβάνει τη βία στους δρόμους. Στις 10 Οκτωβρίου Υπήρξαμε μάρτυρες αυτού κατά τη διάρκεια του Gay Parade και του ποδοσφαιρικού αγώνα στην ε, Τζένοβα. Αυτοί που βιοπράγησαν ε, κινήθηκαν με πολιτικό τρόπο και έστειλαν κάποια μηνύματα και τα συνθήματα που ακούστηκαν συμπεριλαμβάνοντας αυτό. Αυτή είναι και η σκοτεινή συνέπεια του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Θα πρέπει να δούμε ποιες πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν αυτού του είδους τις πράξεις. Θα πρέπει να απαγορευτούν. Μια δημοκρατική χώρα πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι λυπηρό αυτό που κάνει και η Σερβική Εκκλησία πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα διλήμματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Σερβία και ελπίζω η Σερβία να μπορέσει να κάνει μια κάθαρση από αυτή την κληρονομιά που έχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Atkins πρώτα. Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω. Δεν θα επαναλαμβάνω μέχρι κορεσμού αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Οι παράγραφοι 4 και 5 είναι πολύ σημαντική Συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απαραίτητη και θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και για το κοσυφοπαίδιο. Συγχαίρω τον κύριο Κατσίν για την έκθεσή του, για το ψήφισμά του που είναι πολύ λογική και να συγχαρώ και τον κύριο Σέφλινγκ για την πολύ γλαφυρή και εύγλωτη παρουσίαση των θεμάτων της αστυνομίας, της διαφθοράς και το καθεξής. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ κυρία Μονίθ και μετά κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεση αυτή που μιλάει για την πρόοδο και στις μεταρρυθμίσεις και στην ακύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, το αίτημα ένταξης, απελευθέρωση θεωρήσεων και ανάγκη συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία, το ψήφισμα του, Ευρωπαϊκού, του, του Κοινοβουλίου για τη Σρεμπρένιτσα, το θέμα της Gay Parade, τη διακριτική μεταχείριση βάρος στο Ρωμά κτλ πολύ καλή έκθεση το σχέδιο ψηφίσματος, αλλά η διαφορετική θέση που έχουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου ε, ευνόησε τη φιλοευρωπαϊκή στάση της σερβικής κυβέρνησης αλλά και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το κοινό ψήφισμα στον ΟΗΕ απέναντι στην μονομερή ανακήρυξη της ε, ανεξάρτησης. Μην ξεχνάτε, ότι ήταν ε, μονομερής η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου και θα ήθελα αυτό να αναφέρεται στο ψήφισμα γιατί αναφέρεται έτσι σε όλα τα διεθνή κείμενα. Ήταν μονομερής η ανακήρυξη η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας από πλευράς Κωσυφοπεδίου. Επίσης θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα, να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας που ήταν πολύ θετικά γιατί πραγματικά σηματοδοτούν ένα, ένα βήμα σύγκληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Σερβία. Σας ευχαριστώ κύριο Πέτερλε. Και μετά κυρία Κορνέλισον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κατσίν για την πολύ καλή του έκθεση. Είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ ρεαλιστική. Έδωσε προσοχή σε όλα όσα μπορούν να αποτελέσουν σημεία προόδου και χαίρομαι που η κατάσταση έχει βελτιωθεί μετά τον προηγούμενο γύρο. Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε όλα τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη βάση του μέλλοντος για τη Σερβία και την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία είναι υποψήφια χώρα και όπως και άλλες υποψήφιες χώρες είναι προς συμφέρον της να τα καταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα για να διευκολυνθεί η ενταξιακή τη διαδικασία. Έχουν τη δυνατότητα και την πολιτική βούληση να το κάνουν αυτό, είμαι σίγουρο. Συμφωνώ βέβαια με όλου εκείνου που τόνισαν τη σημασία των καλών σχέσεων με του γείτονέ τη. Προ όλε τι κατευθύνσει θα προσέθετε εγώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλισον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από αυτά που είπε η κυρία Μπράτνερ, θα ήθελα να τονίσω και εγώ δύο στοιχεία. Καταρχάς, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα με τον τρόπο τον, οποίο συμπεριλάβατε το θέμα της, του Gay Pride στην έκθεση. Παραβρέθησα. Συμμετείχα και εγώ με τους διάφορους συμμετέχοντες στο Pride και ήταν σαφές ότι καταρχάς ε, η αστυνομία ήθελε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων και το κατάφερε, κανείς δεν τραυματίστηκε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εκ των υστέρων να διαχωρίσουμε το θέμα του Gay Pride από τη βία που εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για όλους σας φαντάζομαι το ότι έγινε καν το Gay Pride με ασφάλεια, αλλά καθίσταται σαφέ ότι πρέπει πολλά να κάνουν ε, ακόμα οι σερβικέ αρχέ για την αντιμετώπιση των ομάδων αυτών. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω για το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και αυτό συμπεριληφθήσε με πολύ πετυχημένο τρόπο στην έκθεση. Στην απόφαση του Συμβουλίου της προηγούμενης Δευτέρας και τονίστηκε και η σημασία της πλήρους συνεργασίας. Πολύ δικαίως, γιατί χρειάζεται για την σταθερότητα στην περιοχή. πέρα από τα να οριστεί η πλήρη συνεργασία ως προϋπόθεση, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, παρέσχουν, θα παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί η Σερβία. Και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει και στο Βαλιγράδι και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Ε, συζητάμε τη σύσταση ενός ταμείου για την ε, ανάθεση κονδυλίων για εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τα δύο τελευταία χρόνια της ύπαρξης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δεν έχουμε τόσο χρόνο και ο κύριος Μπράμετς ε, προσεκλήθη εδώ στο Κοινοβούλιο να μιλήσει σε εμά. Άρα, ίσω θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μα πει τι θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει, τι παραπάνω πρέπει να γίνει και πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη μπορεί να βοηθήσει και να συνδράμει τη Σερβία στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη στον κύριο Μιρέλ, θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα το συγγητή ανεβλήθηκε για 11 Νοεμβρίου προθεσμία υποβολή τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή ανεβλήθη, παρετάθη για μία μέρα η προθεσμία. Ο κύριος Μιρέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Κάτσεν, για την πάρα πολύ καλή αυτή πρόταση που μας υπέβαλε. Καλώ ορίζουμε ιδιαίτερα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Δευτέρα, Ο επίτροπο Φίλε ανέφερε με σαφήνεια ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όχι μόνο για τις σχέσεις με τη Σερβία, αλλά προφανώς και για τις σχέσεις με την υπόλοιπη περιφέρεια και την ε, ε, σταθερότητα στην περιοχή, για το ICTY, για το Εθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Κυκλαβία. Είναι σαφή η στάση και του Επιτρόπου Φιούλε. Υπάρχει αυτή η αιρεσιμότητα και είναι πραγματικά πολύ απαραίτητος αυτός ο ούρος. Ωστόσο, τα συμπεράσματα δεν φτάνουν να αναφέρουν ότι η πλήρη συνεργασία ε, εξισώνεται με την ε, σύλληψη, γιατί αυτό ίσως να ερμηνεύει πολύ στενά αυτόν τον όρο. Γιατί ακόμα και αν γίνουν οι συλλήψεις που είναι απαραίτητες και πάλι και περαιτέρω θα χρειαστεί, και περαιτέρω συνεργασία. Ως τώρα η πλήρη συνεργασία είναι ένα θέμα μέσου, όχι αποτελέσματος. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την πρόταση του κύριου Κάτσιν και καλώς την πολιτική απόφαση για να γίνει αυτός ο εκ νέου διορισμός των ε, δικαστών και των εισαγγελέων. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη διαδικασία. Η διαδικασία δεν είναι διαφανής και μπορεί να έχει πολιτικό χαρακτήρα, όπως ε, σωστά σημείωσε ο συνάδελφος Κάτσιν το θέμα του άρθρου 12 των λευκών ε, εντολών. Εμείς θα θέλαμε να ενισχυθεί η διατύπωση. Πρόκειται για ένα τελείως αντιδημοκρατικό σύστημα. Αν απλά επιστήσουμε την προσοχή σε αυτό, ίσως το μήνυμα που αποστέλουμε δεν είναι αρκετά δυνατό. Καλώς ορίζουμε το άρθρο 4 σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό στο σημείο αυτό η Σερβία μπλοκάρει το κωσυφοπαίδιο γιατί δεν αποδέχεται τα τελωνιακά στοιχεία. που είναι απόλυτα συμβατό με την 1244. Ε, Αυτό αποτελεί εμπόδιο για την ε, συμφωνία ΣΕΦΤΑ σε ό,τι αφορά το άρθρο 18 το καλωσορίζουμε, αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο είναι ουσιώδες, θεωρούμε, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ρωμά έχουν έγγραφα ταυτοποίησης, τα οποία δυστυχώς ως τώρα ε, δεν ε, συμβαίνει. Για το άρθρο 24 για τις συμφωνίες έκδοσης, θεωρούμε ότι οι συμφωνίες έκδοσης με την Κορέα δεν συμπεριλαμβάνουν τα εγκλήματα πολέμου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι συμφωνίες, αλλά για την ε, Κροατία δεν συμπεριλαμβάνεται ε, τα κλίματα πολέμου. Δυστυχώς, για να σας γλιτώσω και λίγο χρόνο, Πρόεδρε, θα προτείνω το εξής. Έχω κάποιες ε, ίσονος σημασίας παρατηρήσεις, τις οποίες θα τις διαβιβάσουμε κατηδίαν στον κύριο Κάτσιν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κατσίν έχει τελευταίος το λόγο για τις τελευταίες του παρατηρήσεις, τελευταία του σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρεμβάσεις, συστάσεις, υπενθυμίσεις και ανακοινώσεις και υποβολή τροπολογιών που μπορούν να συμβάλλουν τα μάλα σε ένα πλήρες ψήφισμα για τη Σερβία. Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας στα σχόλια του κ. Σεφλίν που είπε ότι οι μυστικές υπηρεσίες ε, αυξάνονται στη Σερβία. Δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι μειώνεται η επιρροή των μυστικών υπηρεσιών, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος ήταν ε, της υπηρεσίας, ο υπουργός εσωτερικών ήταν εκεί, αλλά ήταν και πρώην διευθυντής της ΜΠΙΑ, της Μυστικών Υπηρεσιών, ε, που εμπόδιζε τη σύλληψη του Μλάντιτς όταν διώχθηκε από τα καθήκοντά του ο δόκτωρ Ντάβιτς όπως αποκαλείται εμφανίστηκε ο κύριος Κάρατζιτς η μυστική υπηρεσία ήξερε πού βρισκόταν αυτός αυτό το μήνυμα από το Βελιγράδι δεν ήταν πολύ θετικό δηλαδή από τη μια πλευρά μειώνεται ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών ταυτόχρονα όμως διαδίδονται κάποια λανθασμένα μηνύματα. Αυτό θα πρέπει να το φροντίσει η Σερβία. Διότι ο εισαγγελέα για την κλίματα πολέμου Βούτσεβιτς κατηγορούσε αυτό συγκεκριμένο άτομο που ήταν υπεύθυνο για ανεπιτυχείς προσπάθειες να συλληφθεί ο Μλάντιτς κατά το παρελθόν. Αναφέρθηκε το 2006 και το 2008. Όσον αφορά κάποιες παρατηρήσεις Τη κυρία Κοπά, τη συγκεκριμένη συναδέλφου κυρία Κοπά, εν πάση περιπτώσει θα υπάρξουν τροπολογίες. Η προθεσμία από την πλευρά μου μπορεί να παραταθεί για μία μέρα τουλάχιστον, αν χρειάζεται. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη στις 8 Νοεμβρίου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε έχουμε μία-δύο μέρες. Στο τέλος όμως το... η διαδικασία επικύρωσης ε, της συμφωνίας έχει δρομολογηθεί και θα πρέπει να προτείνω κάποιες προφορικές τροπολογίες πριν εγκρίνουμε το κείμενο στην ε, Ολομέλεια και τι υπάρχουν εξελίξεις και αδίποτε πρόοδος θα πρέπει να ε, εντοπιστεί και να χαιρετιστεί. Της κυρίας Μπραντνερ τα σχόλια. Διάλυση των παραλλήλων δομών στο Κωσυφοπαίδιο. Είμαι επιφορτισμένος με τη Σερβία και όχι με το Κωσυφοπεδίο ούτε με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θα ενδείκνεται κάτι τέτοιο, αποβάλλετε σχετικώ τροπολογίε. Θα το συζητήσουμε του κοιόδη εισηγητέ, να δούμε πω μπορούμε να συμφωνήσουμε επί συμβιβαστικών τροπολογιών για να συμπεριλάβουμε αυτή την αναφορά για να αποφύγουμε κάποια πολιτική παράπλευρη ζημιά. Δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι τι θα διαβάσουν και τι θα καταλάβουν σαν μήνυμά μας οι Σέρβοι. Το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εύγλωτο. Ο κ. Κούκαν, ο κ. Ντανζάν και εγώ και οι τρεις μας ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να στείλουμε κάποια μηνύματα στη Σερβία και ελπίζουμε να έχουμε θετική ανταπόκριση στο εγγύς Όμως υπάρχει κάτι που θέλω να προσθέσω. Πρώτα απ' όλα δεν είπα τίποτα για διαμεσολαβητή αλλά είναι πολύ σημαντικό θεσμός στη Σερβία και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να χαιρετήσουμε αυτά που συμβαίνουν. Ο Διαμασολαβητή ήδη άνοιξε τρία γραφεία στην κοιλάδα του Πρέσοβο, στους τρει δήμους, για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η πρόοδος. Και υπάρχει και κάτι που θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα στο Κοινοβούλιο Όποτε αναφέρω το Βελιγράδι, προσπαθώ να πείσω τους βουλευτές στην Όποτε είμαι στο Βελιγράδι, προσπαθώ να πείσω τους βουλευτέ Στην συνέλευση της Σερβίας να έρθει εδώ. Προσπάθησα να πείσω την πρόεδρο του, του Κοινοβουλίου να έρθει εδώ. Αλλά δεν υπήρχε θετική ανταπόκριση από το γραφείο του Προέδρου του δικού μα, του κ. Μπούζεκ. Γι' αυτό κάλεσα και εκείνον και το γραφείο του να είναι πιο θετική και να ανταποκριθούν άμεσα. Όχι μόνο σε περίπτωση τη Σερβική Εθνοσυνέλευση και τη Προέδρου, αλλά και στην περίπτωση συνελεύσεως τη Βοηβοδίνα και εσδήποτε τοπική κοινότητα που προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο στην ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο και αναγκαίο. Για μια ακόμη φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στη συνεργασία με του σκιώδει συγγητέ για να εξετάσουμε τις τροπολογίες που θα υποβάλλω τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος συνάδελφε κύριε Κάτσιν. Πάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά τη Διαριγωνική Συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα του προϋπολογισμού. Μετά που ετέθησε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, έπρεπε να επανεξεταστεί η διοργανική συμφωνία όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα προπολογισμού. Το Συμφωνίο ΔΕΤΑ τη Νέα Συμφωνία αναφέρεται στη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ και το σχέδιο γνωμοδότησης που εξετάζουμε προσφέρει μια ανάλυση και ενδελεχή συζήτηση και παρουσίαση του θέματος. Σχεδόν όλες οι διατάξεις παλιάς συμφωνίας, της διοργανικής συμφωνίας, διατηρήθησαν στο κείμενο της νέας συμφωνίας και εισήχθησαν μόνο κάποιες προσαρμογές κυρίως τεχνικής ε, φύσεως. Θέλουμε να δούμε πιο ουσιαστικέ τροποποίησεις σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και σύμφωνα με τη δήλωση για την πολιτική ευθύνη που έκανε η κυρία Άστον. Δίνω το λόγο στην κυρία Μούνιθ, την εισηγήτρια, για να αναφερθεί στις τροπολογίες που προτάθηκαν και να ενημερώσει την Επιτροπή όσον αφορά τους συμβιβασμούς, εκεί που επετέφθη συμφωνία με τους κοιόδης εισηγητές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπω είπατε, η ισχύουσα διοργανική συμφωνία για θέματα συνεργασίας δημοσιονομικής ανάγεται στο 2006. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωσή τη, επικαιροποίησή τη για να προσαρμοστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας και ιδιαίτερα στο άρθρο 36 που είναι αυτό που μας πειράζει περισσότερο και μιλά για την υποχρέωση της ΥΠΑ εκπροσώπου να διαβουλεύεται τακτικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, τα, για τις βασικές πτυχές και επιλογές της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Παρά την απαραίτητη αυτή ουσιαστική προσαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας, η τροπολογία που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περίεχε πολιτικές θέσεις ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά περιοριζόταν σε τεχνικές αλλαγές της δημοσιονομικής διαδικασίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό στην αρχική μου γνωμοδότηση κατέθεσα εννέα τροπολογίες και μία σειρά προτάσεων που μιλούσαν για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και τη λήψη υπόψη των πολιτικών προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αποστολές ε, της ΚΕΠΑ που είχαν κάποιες ε, δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά και την εντολή και την εκτέλεσή τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δίνεται εγκαίρως, εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Και για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις αποστολές να τακτικές συμβουλευτικές ε, συνεδριάσεις ε, ανάλογα με τις πολιτικές αναγκαιότητες πέραν των έξι επίσημων ε, de facto προγραμματισμένων συνεδριάσεων. Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες από την Επιτροπή Επιτροπή, Πολιτικής Επιτροπής Ασφάλειας πριν την συνεδρίαση. Άλλωστε και στην Πολιτική Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν μέλη του Διευρυμένου Προεδρίου των Επιτροπών Εξωτερικών και Προϋπολογισμών, καθώς και οι συγητές ε, και τα ενδιαφερόμενα μέλη, οι αρμόδιοι, οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων σε αυτές τις συνεδριάσεις. Επίσης, προτείναμε ε, κατανομή των διαφόρων ε, δαπανών, των διοικητικών και των επιχειρησιακών, ώστε να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να διενεργήσουμε τον κοινοβουλευτικό δημοσιονομικό έλεγχο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Διευρύναμε τον κατάλογο των δράσεων της ε, ΚΕΠΑ που θα πρέπει ρητά να αναφέρονται στον προπολογισμό, αφήνοντα ανοιχτή και την ε, δυνατότητα να δούμε και κάποιες ε, εξωτερικές δράσεις που δεν περιλαμβάνονται και ρητά. Εκτός από τις 9 αρχικές τροπολογίες που είχα καταθέσει ως συγγήτρια, έλαβα και άλλες 15 περίπου τροπολογίες από τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Με τους κοιόδες συγγητές καταρτήσαμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες που κατά τη γνώμη μου καλύπτουν όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η συμβαστική τροπολογία 1 μιλάει για το διαχωρισμό επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών. Η συμβαστική τροπολογία 2 μιλάει για τις δημοσιονομικές γραμμές που θα πρέπει ρητά να περιλαμβάνονται στο σχετικό κεφάλαιο της ΚΕΠΑ του προϋπολογισμού. Η συμβαστική τροπολογία 3 μιλά για τη σύνθεση και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της ε, Πολιτικής Επιτροπής και Πολιτικής Ασφάλειας που θέλουμε να είναι ε, συνεδριάσεις ε, διαφανής, ε, με ευρύ σύνθεση, φυσικά διασφαλίζοντας ε, την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. Δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλη αυτή η Επιτροπή, δεν θα μπορεί να συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές, αλλά τουλάχιστον τα μέλη του Διευρυμένου Προεδρείου, οι συγητές και οι αρμόδιοι της κάθε ομάδας για τα συγκεκριμένα θέματα. Να εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολιτικές ομάδες, γιατί δεν έχουν όλες οι πολιτικές ομάδες συγητές για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και μηχανισμούς της εξωτερικής πολιτικής και η τέταρτη συμβαστική λύση αναφέρεται στην ανάγκη ενημέρωσης ε, της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ε, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αυτών των ε, αποστολών και δράσεων της κοινή εξωτερικής πολιτικής. Ευελπιστώ ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα ικανοποιήσουν τις πολιτικές ομάδες και τους συντάκτες των υπόλοιπων τροπολογιών γιατί θεωρώ ότι το πνεύμα τους τουλάχιστον καλύπτεται και ελπίζω να καταρτήσουμε και ένα κατάλογο ψηφοφορίας που θα ικανοποιεί το σύνολο των βουλευτών. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μονίθ για αυτή την γνωμοδότηση. Είναι πολύ σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο εν ώψη της συζητήσης στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ήθελα να επιθυμίσω δύο αλληλένδετα στοιχεία. Η αλλαγή της δομής του προπολογισμού της ΚΕΠΑ δεν είναι μόνο κάτι τεχνικό, αλλά και πολιτικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάτι που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έχει σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά μια διάσταση της εξωτερικής δράσης της Ευρώπης κάτι που ανέθεσε μέσω διακυβερνητικής προσέγγισης η συνθήκη όσον αφορά τις λήψεις αποφάσεις, λήψη αποφάσεων και όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ε, να εξαλειφθούν οι υπερβολές που εμπεριείχε η πλήρη συναπόφαση και να μπορεί το Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του όσον αφορά τον προπολογισμό και όσον αφορά την ΚΕΠΑ είναι πάρα πολύ αποφασιστικό. Και πρέπει να ληφθεί και κάτι άλλο υπόψη. Στην έγκριση του δημοσιονομικού κανονισμού αυτή η αρχή συμπεριλήφθη άμεσα στην πρωτογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γιατί ο δημοσιονομικός κανονισμός δέχτηκε το Συμβούλιο δέχτηκε τη θέση μας όσον αφορά το θέμα αυτό, οπότε ο δημοσιονομικός κανονισμός ήδη ενστερνίζεται αυτή την αρχή ότι τουλάχιστον οι τρεις σημαντικές αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να έχουν ξεχωριστά κονδύλια από τον προπολογισμό. Και αυτό συνδέεται με το δεύτερο θέμα που καλύπτεται σωστά στη γνωμοδότηση, το μεγαλύτερο βάρος στα Joint Consultation Meetings γίνονται meetings που δεν αντιμετωπίζουν μόνο θέματα προπολογισμού, τεχνικά θέματα, αλλά και πολιτικά ζητήματα. Και συνεπώ η παρούσα συμμετοχή, που είναι κυρίω ο πλευρά τη Επιτροπή Προπολογισμών. Εγώ είμαι μόνιμο εισηγητή για τον προπολογισμό τη ΚΕΠΑ στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είναι μείωση όμω, ήταν μειωμένη η εκπροσώπηση τη ΑΦΕΤ και αλλάζει αυτό διότι εκεί υπάρχει κάλυψη και από πλευράς του υπολογισμού και από πλευράς πολιτικής. Και γι' αυτό έκανα, γίνεται αυτή η πρόταση του συμβιβαστική τροπολογίας. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράτνερ, έχει το λόγο. Σκιώδης εισηγήτρια των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ το συντάχτη για, το, για την πρόταση ψηφίσματο. Ήταν πολύ καλή συνεργασία, τον ευχαριστώ. Είναι κοινή η γραμμή μα όσον αφορά τι πτυχέ και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η γνωμοδότηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα για το Κοινοβούλιο. Και όπω υπογράμμισε και ο συνάδελφο Γκουαλτιέρη, είναι πολιτικό ζήτημα, διότι πραγματικά θα θέσει τι βάσει για τον έλεγχο, το δημοσιονομικό του Κοινοβουλίου και πολιτικό έλεγχο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Οπότε αυτό θα καθορίσει τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια και πόση εξουσία θα έχουμε στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα. Θα πρέπει να εξομαλυνθεί η δημοσιονομική διαδικασία για την ΚΕΠΑ και το ίδιο να γίνει και σε άλλου τομεί πολιτική. Δεν θα πρέπει να ο, περιορίζεται πλέον ο, ο λόγος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προπολογισμό για την εξωτερική πολιτική, όσον αφορά το δημοσιονομικό έλεγχο, είναι καλό που θα έχουμε τα ξεχωριστά κονδύλια, κάτι που αναφέρθηκε για την ΚΕΠΑ και τι σχετικέ αποστολέ, εξωτερικέ δράσει και για του ειδικού εκπροσώπου, διότι έτσι θα μπορούμε να αντιδρούμε και να ελέγχουμε τι αποστολέ πάρα πολύ καλύτερα. Και ελπίζουμε να υπάρχει και διευρυμένη υποβολή αναφορών στο Κοινοβούλιο και ενημέρωση του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε και στο μέλλον ετήσια στρατηγική για την ε, ε, διάδοση της ειρήνης όπου θα καθορίζονται οι στόχοι που επιδιώκονται και τι πόρους χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε θεματικές εκθέσεις ε, που θα αναφέρονται στα διάφορα οικονομικά μέσα, να δούμε τι κάνουμε και έτσι ελπίζουμε ότι θα βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών που ακολουθούμε σε αυτού του τομεί. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση η κυρία Λέζινγκ, που είναι η σκιώδη συζητήτρια τη ΓΚΟΕ. Σα ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Η ομάδα μου και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ε, διαθεσμικέ συμφωνίες, για τη μεγαλύτερη διαφάνεια για τα μεγαλύτερα δικαιώματα ελέγχου του Κοινοβουλίου και συμφωνούμε με τις προτάσεις αυτές. Συμφωνούμε και με τις πιο πολλές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των χρηματοοικονομικών μέσων, εγώ και η ομάδα μου, όπως αναφερθήκαμε, Absolut gegenteiliger Meinung. έχουμε καταθέσει τροπολογίες όπου εκθέτουμε τη θέση μας και δεν νομίζω ότι υπάρχει νομοποίηση για στρατιωτικές ε, επεμβάσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή έστω και ανθρωπογενών καταστροφών. Δεν δικαιολογείται στρατιωτική επέμβαση και δεν θα πρέπει να δίνονται κονδύλια για στρατιωτικοποίηση ή στρατιωτικοποιημένη προστασία των πληθυσμών που έχουν πληγεί από οποιαδήποτε καταστροφή. Διαφωνώ με αυτήν την ιδέα ζήτησε να μιλήσει ο συνάδελφος Αλαφράγκα, τελευταίος μένα, αλλά εξίσου σημαντικό. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπαμε, αυτή είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή προπολογισμών που προσπαθεί να διευκρινίσει το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ΚΕΠΑ και ιδιαίτερα για τη δημοσιονομική διαδικασία της ε, ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνηση από την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα παράτασης πέρα των προβλεπομένων για όλη την περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών που είναι εξαετής τα μη χρησιμοποιημένα κονδύλια, τις μη χρησιμοποιημένες πιστώσεις κατά την τρέχουσα δημοσιονομική χρήση. Γιατί ε, ίσως ε, μπορούμε να μεταθέσουμε τα κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Πολλοί είναι ενθουσιώδεις με αυτή την ιδέα. Εγώ πάντως ε, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο από άποψη δημοσιονομικής τεχνικής να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εξαιτίας. Γιατί είναι πολύ περίπλοκη η δημοσιονομική διαδικασία. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο εκαθάριση λογαριασμών, να δίνεται η απαλλαγή. Μια τέτοια παράταση καθ' όλη τη διάρκεια της εξαιτίας, η δυνατότητα χρήσης των χρησιμοποιητών πιστώσεων ε, μέσα στην εξαιτία, έχω κάποιες αμφιβολίες. Ήθελα να ακούσω και τη γνώμη της συγγήτριας. Επίσης, πριν να δοθεί έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος των δημοσιονομικό γραμμών, θα πρέπει η εκπρόσωπος να λάβει υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ έξυπνο αυτό το στοιχείο για να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να μην έχουν απλώς ρητορικό χαρακτήρα ή διακηρυκτικό χαρακτήρα τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω λάβει ακόμη τις συμβαστικές τροπολογίες που ανέφερε η συγκήτρια. Πριν λοιπόν καταρτήσω τη λίστα ψηφοφορίας για την ομάδα, θα ήθελα να λάβω τις συμβαστικές τροπολογίες για να τις εξετάσω ελεγχώς. Ποια σχόλια της συγκήτριας. Α, μισό λεπτό. Ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον, την εισηγήτρια την κυρία Μονίθ για αυτή την πρότασή της που έχει σαν στόχο την ε, ενίσχυση του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία τη κοινή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο φορέα σε αυτόν τον τομέα. Η διοργανική συμφωνία είναι τριμερή. Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο συμμετέχουν. Πολλέ τροπολογίε που υπευλήθησαν από την εισηγήτρια θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια των τριμερών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη διοργανική συμφωνία. Επιπλέον η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική με το ρόλο της ΥΠΑ, της εκπροσώπου και της αντιπροέδρου που επικουρείται από την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής σας θα αποτελέσει συμβολή στη συζήτηση για μια νέα συμφωνία που αφορά αυτούς τους διαφορετικούς φορείς, κυρίως όσον αφορά τη μορφή των συνεδριάσεων ε, για τη διαβούλευση θα λάβει χώρα. Όσον αφορά το κείμενο, είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε τη δέσμευση της ΥΠΑ της που θέλει να παίξει ενεργό ρόλο όσον αφορά τη νέα διοργανική συμφωνία. Αυτό το είδαμε και στην ε, δήλωσή της για το political accountability. Στην ίδια δήλωση είπα ότι η εκπρόσωπος δεσμεύεται ε, για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον προπολογισμό για την ΚΕΠΑ και όσον αφορά τις μεγάλες αποστολές. Όσον αφορά αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η συγκίτρια προτείνει επανεισαγωγή στη συμφωνία μιας δημοσιονομικής δομής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη δομή που είναι πλέον συνεκτική και αντιστοιχεί στην δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου όσον αφορά τα εξής. Πρώτα απ' όλα μεγαλύτερη διαφάνεια και δεύτερον διατήρηση τη ευελιξία που χρειάζεται όσον αφορά τον προπολογισμό για την ΚΕΠΑ. Η προτινόμενη δομή, αυτή προτείνει ε, την εισηγήτρια απο, αποφεύγει τον παραπλησιασμό των κονδυλίων και εφαρμόζοντα επίσης, επίση εξασφαλίζοντα διαφάνεια στι μεγάλε αποστολέ που απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι του προπολογισμού. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να διαφωνήσει με τι προτινόμενε τροπολογίε που ακολουθούν όσον αφορά την εκ των προτέρων διαβούλευση του Κοινοβούλου, όσον αφορά τι προθέσει μεταφορών εντό κατηγορία ε, δεν λαμβάνει υπόψη τον αναγκαίο ε, ευελιξία για τον προπολογισμό που αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά τις συνθισμένες πρακτικές, όσον αφορά την τρίμηνη έκθεση που θα πρέπει να παραμείνει και να μην γίνει μηνία έκθεση, κάτι που προτείνεται, θα είχαμε έτσι 12 εκθέσεις ε, που είναι υπερβολικό και, και υπενθυμίζει ότι οι εκθέσεις αυτές είναι εσωτερικές του θεσμικού οργάνου θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, διότι ο προπολογισμό τη ΚΕΠΑ που είναι στην κατηγορία 4 δεν χρηματοδοτεί παρά μόνο δράσει επιχειρησιακέ. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια σχόλια. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ θερμά όλους ε, όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται τις, τις ε, που θέλουν να διευκολύνουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να αυξήσουν την διαφάνεια. Γιατί στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες ε, της ε, Λισαβόνας με την αύξηση, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούται πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται εγκαίρω για τι ε, αποφάσει που που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, εμεί θα ψηφίσουμε αύριο για αυτή τη γνωμοδότηση και θα τη διαβιβάσουμε στην αρμόδια κατουσία για το θέμα αυτό που είναι η Επιτροπή Προπολογισμών. Κρίμα που δεν έχουν μοιραστεί οι συμβαστικέ τροπολογίε πάντω. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να... και πολύ πιο απρόσκοπτη συζήτηση αν είχαν μοιραστεί στους συναδέλφους αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες. Είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το θέμα. Ο κύριος Αλαφράνκα ρώτησε για τα κριτήρια που ισχύουν σε περίπτωση ε, μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων και τη δυνατότητα ε, χρησιμοποίηση τους αργότερα, πέραν του νησιν 2. Λόγω της πενιχρότητας των κονδυλίων και της ε, του πολύ σχνού υπολογισμού σε ό,τι αφορά τα περισσότερα, τις περισσότερες γραμμές. Γι' αυτό πρόβλεψε αυτή τη δυνατότητα. Στη σχεδόν απίθανη περίπτωση που περισσέψουν κάποιες πιστώσεις, εγώ πρότεινα αντί να εφαρμόσουμε τον ΙΣΙΝ e 2 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει δυνατότητα παράτασης ε, και κατανομή σε περισσότερα σε, σε ευρύτερη χρονική περίοδο, συγκεκριμένα καθ' όλη τη διάρκεια του πολιετού δημοσιονομικού πλαίσιου. Γι' αυτό και μόνο το λόγο κατέθεσα τη σχετική τροπολογία, κύριε Σαλαφράγκα. Κύριο Σαλαφράνκο νομίζω θέλει να κάνει κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κυρία Μουνίθ. Είχα καταλάβει θαυμάσια το συλλογισμό σας ε, για την πρόταση της Επιτροπής είναι 9 και εσείς προτείνετε παράταση καθ' όλη τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Αλλά η ερώτηση που έκανα δεν ήταν προς την εισηγήτρια, ουσιαστικά ήταν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί καλέσαμε και την Επιτροπή στη συνεδρία και της δώσαμε το λόγο και είπε ποιε τροπολογίες δεν μπορεί να δεχτεί. Φαντάζομαι, μια και δεν περιλήφθηκε σε αυτές που δεν δέχεται, ότι η τροπολογία 1 γίνεται δεκτή. Πάντως από άποψη Δημοσιονομική τεχνική δεν ξέρω αν είναι εφικτή μια τέτοια πρόταση. Ίσως δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση και στην έγκριση των κονδυλίων στα πλαίσια των διαφόρων μηχανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε και τόνισε ποιες τροπολογίες της εισηγήτριας δεν μπορεί να δεχθεί. Άρα φαντάζομαι ότι την τροπολογία 1 τη δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβεί σε μια διευκρίνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν το κατάλαβα ότι πρόκειται περί τροπολογία 1. Εδώ δεν τοποθετηθήκαμε επ' αυτής, διότι ο συνάδελφος Γενική Διευθύνσεω για τον Προπολογισμό, ο κ. Λεβαντόφσκι, και ο κύριος Λεβαντόφσκι είναι υπεύθυνοι για την χρήση του μέσου ευελιξία. Προφανώ μία αναφορά κατά δύο χρόνια θα δώσει περισσότερα χρήματα που θα έχουν κινητοποιηθεί και θα είναι κάτι πιο σημαντικό σε περίπτωση κρίση. Υπενθυμίζω ότι το μέσο ευελιξία θα πρέπει να πληρεί κάποιε ε, όρου για να κινητοποιηθεί. Ε, θα πρέπει να, θα πρέπει να ξεπερνάτε κάποιο, κάποιο όριο κάποιες κατηγορίες. 200 εκατομμύρια το χρόνο στα τρία χρόνια έχουμε 600 εκατομμύρια σαν μάζα. Αυτό επεκτείνεται σε μία περίοδο και αυξάνεται το ποσό και γίνεται δίνεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελίξια για τις διάφορες κατηγορίες του δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά το μέσο ευελιξία δεν αφορά μόνο την κατηγορία 4, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλε τι κατηγορίε του δημοσιονομικού πλαισίου. Το θέμα είναι ευρύτερο και επισέρχεται στην πολύ ευρύτερη συζήτηση τη δημοσιονομική ευελιξία όσον αφορά τι διάφορε κατηγορίε και τα ανώτατα όρια. Δεν θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Αν επιτρέπετε, θέλω να επανέλθω στην εκ των προτέρων ενημέρωση. Εγώ αναφερόμουν μόνο στις μεταφορές των κονδυλίων, κυρία Μουνίθ, όχι στο διάλογο με το Κοινοβούλιο εκ των προτέρων όσον αφορά τι αποφάσει. Όσον αφορά τι μεταφορέ κονδυλίου, ο δημοσιονομικό κανονισμό υπενθυμίζω επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μεταφορέ εντό τη κατηγορία. Το να υπάρχει εκ των προτέρων ενημέρωση σε αυτό το τομέα ε, είναι ενάντια στο δημοσιονομικό κανονισμό και δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος, αλλά πολιτικός πώς δημιουργεί προβλήματα, διότι χρειαζόμαστε να κινηθούμε πολύ γρήγορα καμιά φορά για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις κάνοντας μεταφορές εντός των κατηγοριών, πάρα πολύ γρήγορα να κινηθούμε, κυρίως να φάσεις πληρωμές, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες περιστάσεις, καμιά φορά και σε κάποιες κρίσεις. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατηρήσει την ευελιξία της σε αυτή που προβλέπεται από το δημοσιονομικό κανονισμό. Ειδού και ευχαριστώ ε, κύριε Συγγήτρια και κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει άλλος. Πάμε στο τελευταίο σημείο λοιπόν. Σχέδιο γνωμοδότησης για αφορά τη συγκρότηση μηχανισμού ταχείας αντίδρασης της ευρωπαϊκής Ενώσεως υπευλήθη από την εισηγήτρια την κυρία Βέμπερ στις 5 Οκτωβρίου. Κατετέθησαν 24 τροπολογίες να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θεώρησε ότι δεν μας επέτρεπε ο χρόνος να συμμετάσχει στη δυνάμει του άθρου 50 του κανονισμού η δική μας Επιτροπή στις εργασίες η Προεδρία της ΑΦΕΤ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της διασκέψεως των Προέδρων των Επιτροπών, στον κύριο Λένε, όπου αναφέρει ότι αυτή η κατανομή των ευθυνών δεν μπορεί να προκαθορίσει την ανάθεση, μάλλον την, ε, τις διάφορες ανακοινώσεις που μπορεί να εκδώσει η Επιτροπή. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Βέμπερ, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η ψηφοφορία προβλέπεται για την 5η 28 Οκτωβρίου. Το λόγο έχει η εισηγήτρια, κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε και τα αποτελέσματα των συζητήσεων σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ και την σαφή αναφορά ότι ό,τι συμβεί τώρα δεν θα επηρεάσει την ε, ικανότητα, τη δυνατότητα της Επιτροπής αυτής να αντιδράσει στην απάντηση, στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Γιατί η γνωμοδότηση που θα πρέπει να υποβάλουμε τώρα προς την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν θέλω να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη υπόθηκαν κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να αναφέρω το εξή. Στην Επιτροπή, Ανάπτυξη, στο σχέδιο έκθεση που εκδόθηκε, μία πτυχή που είναι σημαντική και για μας εδώ είναι ότι θα ήθελαν να υπάρχει ένας επίτροπος ο οποίος να είναι αρμόδιος για τις ε, μηχανισμούς ταχείας αντίδρασης. Δεν διευκρινίζεται ποιος. Θεωρώ ότι δικό μας καθήκον είναι, σε εισαγωγικά η λέξη καθήκον, ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει να είναι η... ο ύπατος εκπρόσωπος για τις εξωτερικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Καλωσορίζω την ε, τροπολογία που κατέθεσε λοιπόν ο κύριος Ντανζόν η οποία αναφέρει να δοθεί έντολη στην ύπατη εκπρόσωπο για να δημιουργείται τέτοια μονάδα ταχείας αντίδρασης. Φυσικά και η ομάδα μου και εγώ θα ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας αυτής και προτείνω και οι υπόλοιπε οι ομάδες να την υπερψηφίσουν. Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα για την γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με τη χρήση της πολιτικής ικανότητας αλλά και της στρατιωτικής ικανότητας. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να διευκρινίσω ότι προσπάθησα να είμαι ρεαλίστρια, να ακολουθήσω και την γραμμή που ήδη επικρατεί σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Δήλωσα λοιπόν σαφώς ότι η πρόσβαση τη στρατιωτικής ε, δύναμης θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Αυτό όμως ίσως και να σημαίνει ότι είναι, να είναι η πρώτη λύση που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε δυστυχώς. Να είμαστε όμως και εμ, για τις κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΟΗΕ και επικυρώθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν σαφείς κανόνες για το πώς ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές αυτές δυνάμεις. Δεν μπορώ ασφαλώς να πω ότι δεν πρόκειται να αποδεχτώ τις τροπολογίες που προήλθαν. Επιτρέψτε μου να πω από την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος, γιατί πρόκειται για ιδεολογικό θέμα σε μεγάλο βαθμό. Επιμένω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη και πιο γρήγορη αντίδραση. Δεν λέμε να αποστείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε μια περιοχή κρίσεως, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που έχουμε. Ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή μας να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Και θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Νταουνζά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Ρενάτε Βέμπερ για την εξαιρετική της ε, δουλειά και την πολύ ρεαλιστική της γνωμοδότηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις πολιτικο-στρατιωτικές πτυχές. Υπάρχει το πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη απλώς. Και το είπαμε και από ευκαιρία της ε, συζήτησης Έλντερ. Εγώ είμαι κατά αυτών των ε, ιδεολογικών ε, υποψιών ότι γίνεται εσκεμένα μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης ε, της παρουσίας μας και η χρήση των στρατητικών μέσων είναι η έσχατη λύση. Δυστυχώ όμω πολλέ φορέ, ε, μερικέ φορέ τουλάχιστον, η έσχατη λύση είναι η πρώτη διαθέσιμη λύση, πιο προσιτή για την αντιμετώπιση μια καταστροφή, για τα μεταφορικά μέσα για παράδειγμα. Και κατέθεσα και τροπολογία για τα μέσα μεταφορά, γιατί για τα εναέρια μέσα μεταφορά, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ μακάρι να αλλάξει το μέλλον, αλλά είναι πολύ εξαρτημένη από τα στρατιωτικά μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ ισορροπημένη και ενστερνίζομαι πλήρως τα λεγόμενα της συγγετρίας. Να δώσουμε το λόγο στην αντιπρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο Πάσκου. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και θα ήθελα να υποστηρίξω και την άποψη που εξέφρασε ο κ. Νταουζάν και η εισηγήτρια. Δηλαδή είναι αναπόφευκτο να καταφεύγουμε σε κάποια στρατιωτικά μέσα σε τέτοιες περιστάσεις. Ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι διότι αυτά τα μέσα υπάρχουν. Είναι εκεί. Και αν δεν χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ιδεοδός θα πρέπει να φτάσουμε στην κατάσταση κατά την οποία θα πρέπει την τις πολιτικές και κρατικέ ικανότητε θα πρέπει να τις συνενώσουμε και να αφήσουμε τις στατιωτικέ ε, δυνατότητες στο υψηλότερο κομμάτι του φάσματος, αλλά είναι και θέμα κόστους. Γιατί να επαναλαμβάνω στον πολιτικό τομέα κάτι που ήδη υπάρχει και στο στρατιωτικό τομέα. Και δεν το χρησιμοποιώ το μέσο αυτό γιατί το οδηγούν μόνο ένστολοι. Εκείνοι που φοβούνται ότι οι ένοπλες δυνάμεις, οι ένστολοι, θα έχουν μεγαλύτερο λόγο στην ζωή κάθε χώρας δεν είναι ρεαλιστές. Διότι υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν το όλο θέμα. Η κυρία Μπράντνερ και μετά Λέζινγκ, το επόμενο όνομα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, καλή σας δουλειά κυρία Βέμπερ. Τρία θέματα θέλω να τονίσω. Το ένα θα συζητήθηκε ήδη σε ό,τι αφορά την αντίδραση ε, της στρατιωτική αντίδραση. Όπω είπε και ο προηγούμενο συνάδελφο, είναι η έσχατη λύση αυτή. Κάτι άλλο σημαντικό να διακρίνουμε την ε, αντίδραση στις καταστροφές και την αντίδραση σε κρίσεις. Γιατί υπάρχει αλληλεπικάλυψη, αλλά όχι πάντα και στο πλαίσιο αυτό να κάνω μια προφορική τροποποίηση για την τροπολογία 22 ως εξή τονίζει ότι η αντίδραση στις ε, καταστροφές disaster να διευκρινίσουμε στην ε, τροπολογία 22 ότι μιλάμε για την αντίδραση σε καταστροφές disaster. Είναι σημαντικό αυτό. γιατί δεν μιλάμε για, γενικά, για αντίδραση γενικά σε διάφορες πολιτικές ε, κρίσεις. Κάτι άλλο. Ποιος είναι ο ρόλος ε, της Επιτροπής, της ε, κυρίας Άστον και το καθεξής. Νομίζω ότι για την εφαρμογή της ανθρωπαστικής βοήθειας χρειαζόμαστε την Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συντονισμό με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αν δεν υπάρχει ο συντονισμός αυτός, θα παραμείνει το status quo. Να κάνω προφορική τροπολογία για την τροπολογία 3 ως εξή. Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι άλλο disaster, άλλο crisis. Η εφαρμογή της αντίδρασης των αποφάσεων αντίδρασης σε ε, καταστροφές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανθρωπαστική βοήθεια, θα πρέπει να αποτελέσει βασική αρμοδιότητα αλλά να συμπεριληφθεί και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό ενείται συμβιβασμού μεταξύ της λύσης του κυρίου Νταντζάν και της κυρίας Λούζινγκ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να, να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια. Και θα πρέπει πάντα η ανθρωπιστική βοήθεια να είναι ουδέτερη. Αυτό είναι πάντα αρχή. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ο γενικός συντονιστικός ρόλος του ΟΗΕ, να μην υπάρχει επικάλυψη, να μην αφαιρέσουμε αυτή την αρμοδιότητα από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αλλά να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες του ΟΗΕ. Και θα ήθελα να συζητήσουμε και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόταση της Επιτρόπου Τζορτζέβα. Η ομάδα μας διοργανώνει και σχετική ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες από ενώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και από γερμανικής πλευράς και σας καλώ να συμμετάσχετε σε αυτή την ακρόαση αν θέλετε. Λίγο, κολέγα Συνάδελφος ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Βέμπερ. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κύκλο ανταλλαγής απόψεων, δεν μπορεί να συμφωνήσει η ομάδα μου με την παρούσα διατύπωση, με την παρούσα μορφή του έκθεση και επειδή δεν δεχτήκατε τη τροπολογία μας, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη στάση μας αυτής. Εξέφρασα συχνά ποια είναι η στάση της ομάδας μου για την ε, συνδυασμό πολιτικής και στρατιωτικής ε, ικανότητας. Θεωρώ ότι η χρήση της στρατιωτικής δύναμης ούτε από πλευράς οικονομικής αποδοτικότητας αξίζει τον κόπο, γιατί αν δεν έχουμε ακόμα, αν θέλετε, τις δυνατότητες να επέμβουμε με πολιτικό τρόπο, αυτό οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης το γεγονός ότι η πολιτική αντίδραση δεν είναι επαρκής. Δεν έχουμε αρκετά ελικόπτερα, δεν έχουμε αρκετές υποδομές και αυτό θα επιδεινωθεί γιατί ο κόσμος ε, στον οποίο ζούμε έτσι έχει και, δεν μπορεί, και πρέπει να αλλάξει. Καταλαβαίνουμε ότι Οι καταστροφές προαπαιτούν την χρήση των αξιο... την αξιοποίηση των απαραίτητων πόρων, πολιτικών πόρων, για να μπορέσουμε να αντιδρούμε με αποτελεσματικό τρόπο στις κρίσεις αυτές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω προσωπική παρατήρηση, διότι έχω κάποια εμπειρία όσον αφορά τέτοια προγράμματα συνεργασίας Συμμερίζομαι τις τοποθετήσεις του κυρίου Ντανζάν και του κυρίου Πασκού αλλά σε το, το να εξορθολογήσουμε το κόστος είναι απαραίτητο πολιτικά, κυρίως στιγμές που περνάμε χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες και η διεθνής κοινότητα. Δεύτερο, τα στρατιωτικά μέσα πολύ συχνά είναι πολύ πιο επαρκή και αποτελεσματικά εν συγκρίση με τα πολιτικά μέσα. θετικό μέσα είναι ένα εργαλείο εντελώς ουδέτερο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο ανάλογα με την ανάγκη. Τελευταίο σημείο. Δεν θα, με σκανδαλιζόμουν από το ότι χρησιμοποιούνται ακόμα όχι θετικά μέσα αλλά και ε, ένστολοι σε παρέμβαση κατά φυσικών καταστροφών. Όποιο έχει εμπειρία από παρεμβάσει σε τέτοιε περιπτώσεις, καμιά φορά για να είναι αποτελεσματική και δυνατή η χορήγηση βοηθείας, χρειάζεται Χρειάζονται άντρε, χρειάζονται ένστολοι δυνάμει τη τάξη, στρατιωτικέ δυνάμει που εγγυώνται την τάξη και την ε, ασφάλεια των ατόμων που παρεμβαίνουν, ε, των εκπροσώπων των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Εγώ δεν βρίσκω ε, κάτι κακό θα χρησιμοποιούνται είτε στατιωτικές δυνάμεις είτε στατιωτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει καταρχάς την ε, ομάδα, λέει ο μιλητής, για την προσοχή που προσδίδει σε αυτό το θέμα. Όπως είπε και κάποιος ο μιλητής Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις χτες, υπέβαλε μια ανακοίνωση όπου εκεί αναφέρονται διάφορες προτάσεις για πολιτική για να αναπτυχθεί η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται σε καταστροφές. Αυτή η ανακοίνωση προτάθηκε χτες και ήταν πρωτοβουλία της Επιτρόπου Τζόρτζεβα που είναι υπεύθυνη για την αστική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα βρείτε σε αυτή την ανακοίνωση διάφορες προτάσεις οι οποίες ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση όπως και αρχική έκθεση και απηχούνται και στη γνωμοδότηση της ε, ομάδας. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση και τις υποβληθήσεις και συζητούμενες τροπολογίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την ισορροπία που, που δημιουργούν οι συνθήκες όσον αφορά τους θεσμικούς ρόλους και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μια και της ΥΠΑ της εκπροσώπου από την άλλη, και εδώ αναφέρομαι στην τροπολογία υπαριθμών 2, η οποία κατά την άποψή μας πηγαίνει πολύ μακριά προς κάποια κατεύθυνση και πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς την ισορροπία που προσεκτικά καθορίζεται από τη συνθήκη. Τα άρθρα 196 και 214 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθιστούν σαφέστατο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία η πολιτική, που είναι τα δύο βασικά μέσα με τα οποία ανταποκρίνεται σε κατεπίγουσες καταστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επ' αυτής της υποθέσεως εργαζόμεθα. Στην ανακοίνωση λοιπόν που υποβάλαμε εχθές θα βρείτε μεταξύ άλλων και πρόταση για τη δημιουργία μονάδας ε, ταχείας αντιδράσεως ε, που θα συναθρίζει το σύστημα ε, την αίθουσα για την αντιμετώπιση των κρίσεων και το ΜΙΚ, το μέσο, και θα υπάρχει εστιακό σημείο εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλε τι ε, δράσει για αντιμετώπιση κατεπηγουσών καταστάσεων. Και η ανακοίνωσή μα λέει ότι αυτό το εστιακό σημείο θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω, βεβαίω, βεβαίω. Και θα πρέπει να υπάρχει και πολύ στενό συντονισμό μεταξύ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι εντό εντολή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρω στην γνωμοδότηση κατά την άποψή μου. Πιστεύουμε ότι ένα, κάποια σύγχυση δημιουργείται και από την ορολογία. Πιθανότατα θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι κατά πόσο αναφερόμαστε σε αυτή τη γνωμοδότηση σε αντίδραση σε καταστροφές ή σε διαχείριση κρίσεων και νομίζω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη διάκριση που πρέπει να γίνει σε καταστροφέ ανταποκρινόμαστε καταρχά με ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια όσον αφορά την πολιτική προστασία. Σε κάποιε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει υπάρχει και ανάγκη να έχουμε και εργαλεία αντιμετωπίσεω κρίσεων. Αλλά αυτό είναι σε πολύ ειδικέ περιπτώσει και μόνο. Η πρώτη αντίδραση σε σεισμού, πλημμύρε, σε όλα τα είδη φυσικών καταστροφών είναι μέσω παροχή ανθρωπιστική βοηθεία ή ε, αρρωγή όσον αφορά την πολιτική προστασία. Στην τροπολογία 2 αυτή είναι η απάντηση. Ίσως θα ήταν καλύτερο να αναφερόμαστε σε διαχείριση κρίσεων αντί αντίδραση σε καταστροφές. Και αν δημιουργηθεί ομάδα κρούση task force για να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις, τότε προφανώς στο βαθμό που αυτό καλύπτει αντιδράσει σε καταστροφές θα πρέπει να είναι μεικτή ομάδα κρούση που καλύπτει και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις άλλες αρμοδιότητες. Όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα, Θέλω και εκεί να είμαι ξεκάθαρος, ηλίου φαϊνότερος. Βλέπουμε ότι οι στατιωτικές δυνάμεις, στατιωτικά μέσα μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα ανταποκρινόμενα σε καταστροφές. Αυτό δεν το αρνούμεθα. Αναγνωρίζουμε σαφώς αυτό το θέμα και στην ανακοινωσή μας στατιωτικά μέσα μπορούν να είναι πολύτιμη, πραγματικά πολύτιμη υποστήριξη όσον αφορά τους φορείς πολιτικής προστασίας που ανταποκρίνονται σε καταπήγωσης καταστάσεις, είτε παρέχοντας επιμελητία, μεταφορές ή διάφορα μέσα συγκεκριμένων αντιδράσεων. Υπάρχουν κάποιες ειδικέ περιπτώσεις όπου στερετικά μέσα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση σε μεγάλες καταστροφές. Όμως οι κανόνες και το πλαίσιο για όλα αυτά είναι εξίσου σαφή καταρχήν είναι, χρησιμοποιούνται μόνο σαν τελευταίο μέσο και αυτό αναφέρεται ρητά στην Ευρωπαϊκή Συνένεση που αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε πολύ ε, σημαντικά προβλήματα μπορεί γρήγορα να είναι έσχατη ανάγκη τα στρατιωτικά μέσα και υπάρχει χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν εξ αρχή, διότι η κλίμακα είναι τέτοια τη καταστροφή που χρειάζεται από την αρχή να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικά μέσα. Ο κανόνα και η αρχή είναι σαν έσχατο μέσο χρησιμοποιούνται τα στρατιωτικά μέσα. Η ανακοίνωσή μας αναγνωρίζει ότι τα θετικά μέσα μπορεί να δραματίσουν χρήσιμο ρόλο και επίσης αναφέρεται ότι θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για το συντονισμό μεταξύ της, εξωτερικής, της, ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως και των θετικών μέσων θα υποβληθούν από πλευρά είπα τη Εκπροσώπου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένες προτάσεις. Στην τροπολογία 7 συγκεκριμένα, Πρόεδρος, παρακαλώ αν μπορείτε να ολοκληρώσετε σχετικά γρήγορα διότι μας τελείωσε ο χρόνος. Μάλιστα, πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τροπολογία 7 γίνεται λόγος στις ε, μονάδες μάχης, battle groups, η εντολή τα μέσα και οι στόχοι αυτών των battle groups είναι πολύ διαφορετικοί στόχοι από ό,τι για ανταπόκριση σε καταστροφές σήμερα, οπότε πιθανότατα δεν είναι το σωστό μέσο για να χρησιμοποιηθεί για κάποια αντίδραση σε καταστροφές, εκτός αν γίνουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις εντολές που τους δίνονται και τέλος στην τροπολογία 13 γίνεται αναφορά στην ε, πολιτική άμυνα σαν έσχατο μέσο ε, και εκεί αυτό δεν αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Συνένεση και η πρότασή μας θα ήταν απλώς να κρατήσουμε την διατύπωση στην οποία συνεφώνησαν τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτά είναι όσα είχα να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σύντομο σχόλιο στην εισηγήτρια. Πολύ σύντομα λέει η συγκήτρια. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ των προτέρων. Σε αυτή τη φάση ποια είναι η κατάσταση και διακόπτω το μικρόφωνο της συγκήτριας. Θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με το τι θέλουμε να ληφθεί υπόψη και τότε όταν θα συζητηθεί ελπίζουμε η ανακοίνωση η ΑΦΕΤ θα είναι η καθήλια αρμόδια, ελπίζουμε. Θα ξαναρχίσουμε την όλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι για την ώρα θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να σας πω ότι κάποια από τα θέματα τα οποία εφήγησαν από τους συναδέλφους των Πρασίνων καλύπτονται από την έκθεση της ΔΕΒΕ καθίσταται σαφές ότι αφορά φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντανζάν, για ένα τάχιστο σχόλιο, πάρα πολύ γρήγορο, διότι δύο θέματα εθίγησαν που αφορούσαν τις τροπολογίες μου πρώτα απ' όλα. Ξέρω τι είναι η διαχείριση της κρίσης και τι γίνεται με τις φυσικές καταστροφές. Ξέρω ότι έχουν νόημα οι λέξεις και ξέρω ότι η πραγματικότητα κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Τι διαπιστώνω. Ξέρω τη διαφορά, έλεγα, μεταξύ διαχειρήσεως κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Ε, οι λέξεις έχουν μια έννοια και μια πραγματικότητα που κρύβεται από πίσω έχει διαφορά. Εγώ γιατί είπε την τροπολογία 2, ότι έχουμε κάποια μέσα για αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων, ε, όπως είναι στην ΑΕΤ, χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβουλίου, μπορούμε να μιλήσουμε για καλύτερη συνεργασία, καλύτερο συντονισμό, αλλά εγώ θα ήθελα αυτά να λειτουργούν πιο γρήγορα και καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Αυτό που μετράει είναι αποτελεσματικότητα για μένα και νομίζω ότι η εντολή που δίδεται στην ύπατη εκπρόσωπο είναι ένα πλαίσιο αποτελεσματικό της χρήση των μέσων. Μετά για τα battle groups καταλαβαίνω τους αντιρρήσεις σας. Έχετε δίκιο νομικός όσον αφορά αυτό που θέτετε. Εγώ έχω πολιτικό θέμα και εδώ πολιτικό θέμα προβάλλουμε. Επανειλημμένα σε διάφορα βήματα ζητήσαμε η εντολή των battle groups να προσαρμοστεί ούτως ώστε να χρησιμοποιείται με πιο ευέλικτο τρόπο. Από αυτή την έποψη είναι ένα θέμα πολιτικό και Επ' αυτού πρέπει να τοποθετηθούμε. Συμμερίζομαι απόλυτα την απόψή σα. Ευχαριστώ. Στο επανειδήν, λέει ο Πρόεδρο. Καλή σα όρεξη. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία.